Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ και θέλω να σας ζητήσω την προσοχή σας. Σας καλωσορίζω και θέλω να καλωσορίσω εδώ τον ειδικό προσκεκλημένο μας, τον κύριο Hans από το Κέντρο Δημοκρατικού Ελέγχου Ανοπλών Δυνάμων της Γενέβης και τον καθηγητή Μάρτιν Στάνεν του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. Πριν να προχωρήσουμε στα σημεία που αφορούν τις παρεμβάσεις των προσκεκλημένων μας, να θεωρήσω ως δεδομένο ότι θεωρούμε ότι, ότι εγκρίνουμε με συγχωρείτε την ημερησία διάταξη αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, επομένω εγκρίνεται η μερική διάταξη και να προχωρήσω απευθείας στις ακολουθές ανακοινώσει. Εγκρίνουμε τη σύσταση των συντονιστών να διορίσουμε στου ηγητέ τους εξής. Τον κύριο Κυριάκο Τρενταφυλλίδη για την ε, έκθεση Καλίνιγκραντ, την κυρία Ελέν Φλότρο για την συνέχιση της δραστηριότητας TDIP, τον κύριο Κάρλος Κοέλιο, για την έκθεση σε ό,τι αφορά τη σύσταση ενό μηχανισμού παρακολούθηση και αξιολόγηση ε, για την αξιολόγηση τη εφαρμογή του κεκτημένου Σέγγεν. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνονται οι προτάσει αυτέ. Και επίση, παρακαλώ. Κύριε ένα λεπτό να φέρω στα ακουστικά μου. Ευχαριστώ για το θέμα των εισηγητών έχω μια ερώτηση. Έχω μια ερώτηση σε σχέση με τη διαφάνεια της διαδικασίας, γιατί δεν είναι σαφές για μένα σε σχέση με το πώς ε, κάποια μέλη ε, το μη φτυγμισμένο μπορούν να γίνουν εισηγητές. Υπάρχει ένα νέος κανόνας ε, που συζητήθηκε στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων Δηλαδή σε σχέση με το αν θα επιτρέπονται να είναι συντονιστές ε, τα μέλη αυτά. Δεν ξέρω τελικά τι αποφασίστηκε και δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα. Δεν ξέρω τι θα γίνει όταν γίνεται εισηγητής ένα μέλος του Κοινοβουλίου που είναι στην ομάδα των... Ε, στην Ναι. Από ό,τι ξέρω, εμείς ακολουθούμε τους κανόνες που έχουμε από την αρχή της θητείας και έχουν επικυρωθεί αυτοί οι κανόνες από τη συζήτηση στη διάσκεψη των Προέδρων. Συζητήθηκε αυτό το θέμα γιατί αναφέρθηκαν διάφορες εμπειρίες, αλλά... Οι κανόνες ε, που έχουμε τώρα συμπίπτουν ε, απόλυτα με το μοντέλο που ακολουθούμε μέχρι σήμερα και φυσικά να τίθεται κάθε έκθεση για τη συνεδρίαση των συντονιστών μετά από τις διαπραγματεύσεις. Ε, ακολουθούμε πάντα τις συνήθεις διαδικασίες ε, και αν όχι ακολουθούμε το point system. Will you compliment? No, it's exactly what you have just said. I mean, that, that is the way it is. We can send in writing. We, we, we, we can communicate them on, the, Αν θέλετε μπορούμε να σας ε, το γνωστοποιήσουμε γραπτός. Ναι, σας ευχαριστώ. Έχω και άλλη μια συγκεκριμένη ερώτηση. Μιλήσατε για το The System, για το σύστημα αυτό με τους πόντους. Όμως, ε, εγώ μπόρεσα να δω ένα πίνακα όπου έχετε κάποιους βαθμούς ανά ομάδα. Και πώς ακριβώς λειτουργεί ακριβώς αυτό το point system. Κοιτάξτε, ακριβώς εδώ έγκυται το ζήτημα. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι μία εγγεγραμμένος, δεν σημαίνει ότι είναι δεύτερης κατηγορίας ε, μέλος αυτού του κοινοβουλίου. Έχει πλήρη δικαιώματα. Κάποιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων φυσικά είναι για να συμμετέχουν οι πολιτικές ομάδες και τα μέλη που δεν ε, έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη δομή ως ε, μέλη του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ε, περιμένουν να εφαρμοστούν όλα τα δικαιώματα τους και τα καθήκοντά τους ως μη εγγεγραμμένοι γιατί ορισμένοι τρόποι δράσεις ε, εντό του Κοινοβουλίου είναι σχεδιασμένη για τα μέλη των ε, πολιτικών ομάδων. Και όσοι έχουν κάνει την επιλογή να μην έχουν εγγραφεί σε κάποια συγκεκριμένη πολιτική ομάδα, θα πρέπει και αυτοί να πληρούν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, γιατί ισχύει για αυτούς κάποιο ειδικό καθεστώς. Παρακαλώ. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Αλλά νομίζω ότι έχει δίκιο ο κύριο Κλάς. Ε, έχει εκλεγεί. Εγώ μπορεί να διαφωνώ προσωπικά με το πολιτικό του πρόγραμμα, αλλά έχει πει όλα τα ίδια δικαιώματα με τα υπόλοιπα μέλη και ε, εγώ όπω γνωρίζω στην άλλη επιτροπή όπου είμαι μέλος επιτρέπει στους μη γεγραμμένους να συντάξουν εκθέσεις. Ε, ε δηλαδή ε, δεν ξέρω αν πρέπει, το χάρη, κάποιο να ψηφίσει ε, οπωσδήποτε για κάποιον που είναι πολιτική ομάδα, γιατί διαφορετικά ο δικό εκπρόσωπο δεν μπορεί να συμμετάσχει. Κοιτάξτε, μη διεκραμμένοι θα μπορούν να συντάξουν και να έχουν έκθεση και στη ΛΥΜΠΕ. Έχουν γνωμοδοτήσει και στη ΛΥΜΠΕ σύμφωνα με το σύστημα ΤΕΟΝΤ στην Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων ζητήθηκε να δώσει μια γενική ερμηνεία. Αυτή η ερμηνεία υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια και ήδη έχουμε κάνει μια έρευνα και στις άλλες επιτροπές. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν την ίδια προσέγγιση. Θα το στείλουμε γραπτός αυτό σε όλα τα μέλη. We are now ready to Μπορούμε να προχωρήσουμε. Έλεγα ότι ενημερωθήκαμε ότι ο Υπουργό Μίλλερ που αναμενόταν αύριο στην Επιτροπή Λίμπε δεν ε, θα καταφέρει να παρευρεθεί. Έτσι λοιπόν θα, θα έρθει ο κύριος ε, Πιότρε Στάσανσισκ ε, που είναι αρμόδιος για θέματα ασύλου γύρω στις 11.30. Έτσι λοιπόν τροποποιήθηκε ελαφρώς σήμερα η διάταξη ως εξής. Από τις 10 και 10 μέχρι τις 11 θα έχουμε την έκθεση Βέλτ για την, τα PNR Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυστραλίας και από τις 11 στις 11.30 θα ψηφίσουμε για την έκθεση του κυρίου Μούλτερ σε σχέση με ε, της Πρόεδρου για τα κρατικά κατόπιν στις 11.30 θα έρθει ο Υφυπουργό ε, για το, το για το άσυλο και από τις 12 στις 12.30 θα έχουμε μία κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΦΕΜ για να ψηφίσουμε για την έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασία. Παρακαλώ. Ένα αίτημα. Γιατί με ενημέρωσαν ότι μπήκε το σημείο που με αφορά στις 10 και 10 για αύριο στην μισή διαταξή και δεν με ρώτησαν, εμένα δεν με βολεύει και τόσο πολύ. Έτσι λοιπόν είναι δυνατόν να αλλάξουμε με την έκθεση του κ. Δεμέρα και να ξεκινήσω εγώ στις 9 θα ήμουν πιο ικανοποιημένη. We will, we will try to meet your terms, Mrs. Ναι, θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το έτοιμά σα. Έτσι λοιπόν, περνάμε στο σημείο 3, που αφορά την κοινοβουλευτική εποπτεία των Οργανισμών ασφαλεία και Πληροφοριών στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλε μεγάλε δημοκρατικέ χώρε. Στόχο αυτής της ε, αυτό το σημείο να συζητήσουμε εδώ με τους καλεσμένους μας, ε, τον Δ. Χαντς Μπόν από το κέντρο της Γενέβης, το Κέντρο Δημοκρατικού Ελέγχου των Απλών Δυνάμεων και τον καθηγητή Δ. Μάρτιν Τσάνιν του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. Αυτό το σημείο αφορά την εγκαιρεποπτία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με διαβαθμισμένες πληροφορίες. Όλοι γνωρίζετε ότι δεν έχουμε διαπραγματευτεί αυτές τις συμφωνίες με όλους τους φορείς που ε, μπορούν να ε, διαβαθμίζουν ε, τις διάφορες ε, πληροφορίες που αφορούν και τη δική μας εργασία. Επίσης είναι σημαντική μια ισχυρή δυναμική βάση σε σχέση με το πώς διαβαθμίζονται και αποχαρακτηρίζονται οι πληροφορίες. Έτσι λοιπόν θα, διαφωτί, θα έχουμε ενημερώσει για το θέμα αυτό όπιν των μελετών που αναθέσαμε και θα μας ενημερώσουν οι καλεσμένοι μας, ο κύριος Μπόρν. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να παρουσιάσουμε τη μελέτη μας. Είμαστε ευγνώμονες στο, στη Γενική Διεύθυνση του Κοινοβουλίου για, που μας έδωσε την εντολή να αναλάβουμε αυτή τη μελέτη Και ευχαριστούμε επίσης την Επιτροπή σας που μας έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε τη μελέτη αυτή μαζί σας. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε την EUI για τη συνεργασία μας. Γιατί εδώ είχαμε 20 εμπειρογνώμονες το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο. Έχουμε και άλλους συνεργάτες παρόντες εδώ, αν θέλετε μπορούν να απαντήσουν και αυτοί σε τυχόν απορίες. Τώρα θα ήθελα να σας εξηγήσω τους στόχους της μελέτης, τη, τα κύρια συμπεράσματα και τις συστάσεις. Λοιπόν, ο βασικός στόχος της μελέτης είναι να υπάρξει μία εποπτεία της καταστάσεως στα κράτη-μέλη για να εντοπίσουμε τις ε, βέλτιστες πρακτικές και να ενισχύσουμε την εποπτεία του χώρου ελευθερίας, ασφαλείας και ε, δικαιοσύνης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε για το στόχο αυτό έχουμε ε, περιλάβει την Europol, την Eurojust και τη Frontex. Και επιπλέον έχουμε κοιτάξει το CITSEN, δηλαδή το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, ε, σε περίπτωση επιθέσεων κατά τρόπον ώστε να δούμε πώς η εποπτεία μπορεί να σας βοηθήσει και να παρακολουθείτε καλύτερα τις κινήσεις αυτών των οργανισμών. Επιπλέον έχουμε κάνει 40 ή 50 συνεντεύξεις με, στα πλαίσια του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των διαφόρων οργανισμών με 12 ε, μελέτες περιπτώσεων ε, ε, εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και έχουμε προσεγγίσει όλα τα κράτη-μέλη, όλα τα κράτη-μέλη δηλαδή μας έχουν, έχουν ανταποκριθεί. Και τέλος θέλαμε να εξετάσουμε τα, τους οργανισμούς ε, ε, κοινοβουλευτικού ελέγχου για το 2011. Βεβαίως θα αναρωτηθείτε εμένα τι θα μου προσφέρει αυτό, πώς θα μου βοηθήσει να βελτιώσω την εργασία μου και υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους θεωρούμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να εξετάσετε το θέμα αυτό τώρα. Καταρχήν η συνθήκη της ε, Λισαβόνας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της ε, ε, και τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια ζητά να υπάρξει καλύτερη παρακολούθηση της ε, ε, Europol και της Eurojust και επίσης θα πρέπει να υπάρχουν διάφορες λειτουργίες σχετικές με την εσωτερική ασφάλεια που θα πρέπει να παρακολουθούνται και τρίτον και πολύ βασικό Υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με την πρόσβαση πληροφοριών στα πλαίρια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που είναι ε, να συνδεδεμένες με το θέμα αυτό της εποπτείας. Οπότε πρέπει να δούμε πώς τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν το θέμα των διαβαθμισμένων πληροφοριών και να σας παρουσιάσουμε τα πορίσματά μας εδώ. Προτού ε, προχωρήσουμε στην παρουσίαση θα κάνουμε το πρώτο ερώτημα. Πώς διαφοροποιούμε τις, ε, ε, τους οργανισμούς ασφαλείας και εποπτείας διότι δεν έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες. Δεν, ε, οι υπηρεσίες ασφαλείας ε, και συλλογής πληροφοριών ε, δεν μπορούν προφανώς εύκολα να ζητήσουν να παρακολουθήσουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες παραδείγματος χάρη. Οπότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δούμε πώς διεκπεραιώνονται παρεμφερείς εργασίες και αν πρόκειται για διαβαθμισμένες αυτές πληροφορίες πώς αντιμετωπίζονται για να ξέρετε εσείς πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή πώς μπορείτε να χειριστείτε διαβαθμισμένες πληροφορίες, απόρριτες πληροφορίες στα πλαίσια αυτά. Βρήκαμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά αποτελέσματα τα οποία ε, μπορεί να έχουν σχέση με τη δουλειά μας και άλλα τόσα που δεν έχουν σχέση αλλά ε, για να μπορέσουμε να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε εγώ θα παρουσιάσω εδώ συνοπτικά μόνο τα βασικά σημεία. Το πρώτο το οποίο πρέπει να λεχθεί είναι ότι η ανάλυση μας απέδειξε ότι δεν υπάρχει μία μέθοδος η οποία είναι η καλύτερη. Υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει όμως μία κοινή προσέγγιση σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Υπάρχει ένας ε, κοινοβουλευτικός οργανισμός ο οποίος παρακολουθεί και εποπτεύει τους οργανισμούς ε, της πληροφοριών των κρατών μελών. Βλέπουμε λοιπόν ότι και σε κάθε χώρα υπάρχει ένα κοινοβουλευτή, ένας κοινοβουλευτικός οργανισμός και ε, ένα, μια συγκεκριμένη επιτροπή η οποία παρακολουθεί όλες τις υπηρεσίες πληροφοριών. Τώρα, όσον αφορά τον περιορισμό της κοινοβουλευτικής εποπτείας, βλέπουμε ότι στα περισσότερα κράτη, τα κράτη-μέλη δεν ε, εμπλέκονται ε, στο θέμα αυτό της εποπτείας και το αναθέτουν σε ένα γενικό διευθυντή. Ε, και αυτό ήταν ένα σημείο που έπρεπε να αναφέρω. Και τέλος, το τελευταίο που θα ήθελα να σχολιάσω γενικώ είναι ότι οι περισσότερες συμφωνίες ε, ε, μεταδόσεως πληροφοριών ε, μεταξύ εποπτικών οργανισμών και κοινοβουλίων μπορούν να εξεταστούν. Έχουμε δηλαδή ε, πάρα πολλά πορίσματα που αναφέρονται στους οργανισμούς αυτούς, αλλά αυτά τα θέματα ήταν τα πιο βασικά που ήθελα τώρα να τονίσω και να αναφερθώ σε τρία αποτελέσματα σχετικά με την πρόσβαση στις ε, διαβαθμισμένες και απόρριτες πληροφορίες. Το πρώτο είναι ότι οι συνάδελφοί σας στα Εθνικά Κοινοβούλια σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη έχουν ε, πρόσβαση στις απόρριτες απόρριτες πληροφορίες και στις διαβαθμισμένες πληροφορίες. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα κράτος Ευρωπαϊκή Ένωση όπου να αρνούνται εις τους, εις τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Επίσης οι βουλευτές δεν χρειάζεται να ψάχνουν τις πληροφορίες ως επτοπλίστων πρέπει η εκτελεστική εξουσία να συγκεντρώσει τις τις και να τις διοχετεύσει στα εθνικά κοινοβούλια, ιδίως όσον αφορά τα θέματα της εθνικής ασφαλείας. Στα περισσότερα λοιπόν κράτη δεν βλέπουμε να είναι θέμα των των βουλευτών να ψάξουν τις πληροφορίες ε, αλλά πρέπει να τις έχουν εγκαίρως στη διάθεσή τους. Ε, θέλω λοιπόν εδώ να αναφέρω όμως ένα, ε, μία επιφύλαξη ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, για το κατά πόσον μπορούμε να μεταφέρουμε τις εθνικές μεθόδους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή μπορεί να νομίζουμε ότι έχουμε πολλά κοινά στοιχεία με το εθνικό επίπεδο και να δείτε ότι υπάρχουν πολλές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στις ευρωπαϊκές χώρες αλλά παρόλα αυτά πρέπει πάντοτε όλες αυτές οι μέθοδοι να προσαρμόζονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ερχόμαστε τώρα στο τελευταίο μέρος της προτάσεώς μας που είναι οι συστάσεις της παρουσιάσεώς μας που είναι οι συστάσεις και ε, θα ήθελα να πω καταρχήν ότι βάσει των πορισμάτων μας ε, διαπιστώσαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε επίσης να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν περιορισμοί στην εποπτεία αυτών των οργανισμών εθνικής ασφαλείας. Ο πρώτος περιορισμός επί του οποίου θα πρέπει να αποφασίσετε και ε, διαπιστώσαμε από τις εθνικές πρακτικές είναι ότι ε, οποιαδήποτε μέθοδος εποπτείας δεν πρέπει να είναι πολύ ε, περιοριστική και βαριά κατά τρόπον ώστε τα, τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν αυτούς τους οργανισμούς και να συνεργάζονται μαζί τους. Το δεύτερο θέμα που βασίζεται στην εθνική πρακτική και πρέπει να εξετάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι ίσως δεν θα έπρεπε να αναφερθείτε μόνο στη Frontex και στην Eurojust γιατί βλέπουμε ότι στο σε εθνικό επίπεδο τα κοινοβούλια λέγουν ότι άπαξ και αναλάβουμε την διαχείριση αυτών των οργανισμών δεν θα μπορούμε πλέον να τους εποπτεύουμε ανεξάρτητα και θα χρειαστεί ε, κάποια, κάποιο νομοθετικό πλαίσιο που να οριοθετεί τις ε, αρμοδιότητες και ευθύνες αυτές. Και τέλος τέλος διαπιστώσαμε ότι ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βασίζεται ε, όχι τόσο ε, τα βασίζεται λιγότερο στον εαυτό του διότι έχει εποπτικά όργανα που λειτουργούν για, για λογαριασμό του. Είναι πολύ βασικό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, συνεχίσει το διάλογο με ε, τη, τα υποπτικά ε, τους εποπτικούς οργανισμούς που παρακολουθούν την Europol και την Eurojust και θα δώσω τώρα τον λόγο στον συνάδελφό μου για τη συνέχεια. Ευχαριστώ που είσαστε σύντομος και, παρουσιάσατε τον, και παρουσιάζω τον δεύτερο ο μιλητή, τον καθηγητή Μάρτιν Σάινι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ε, πω το εξή ε, ότι ο ρόλος ε, των Οργανισμών Ασφαλείας και Πληροφοριών και σημασία τους έχει αυξηθεί πάρα πολύ από την 11η Σεπτεμβρίου του 2011 όταν οι οργανισμοί ασφάλειας ε, και πληροφοριών ανέλαβαν ε, πάρα πολλά καθήκοντα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, και άλλαξε και το τοπίο, δηλαδή η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των οργανισμών ασφαλείας έγινε πολύ μεγαλύτερη. Στο παρελθόν οι οργανισμοί ασφαλείας και πληροφοριών κατασκόπευαν μία την άλλη, ενώ τώρα στην τρομοκρατία, στο πλαίσιο της τρομοκρατίας βρίσκουν ένα κοινό εχθρό για να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργήσουν παγκόσμιες συμμαχίε. Λεχθέντο αυτού, επίσης ε, συνειδητοποίησαμε ότι σε πολλές χώρες υπήρχε ένα κενό στην ε, νομική ρύθμιση, γιατί ακριβώς ε, θέματα διεθνούς συνεργασίας μεταξύ οργανισμών ασφαλείας δεν είχαν ρυθμιστεί και δεν υπήρχε επαρκής αποπτία. Έτσι λοιπόν, ε, αυτό είναι το background ε, που ήθελα να αναφέρω όταν ήμουν ε, ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της δημοκρατίας. Ξεκινήσαμε την εκπόνηση δύο εκθέσεων για το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΙΕ και το ένα αφορά σε σχέση με τις βαλτικές πρακτικές στην εποπτεία των οργανισμών πληροφοριών και μπορούμε να αναφέρουμε αναφέρουμε ότι πολλά κράτη-μέλη και στην νομοθεσία τους αλλά και στην πράξη κάνουν πολλά πράγματα σωστά και άλλες χώρες θα μπορούσαν να διδαχτούν. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δυνατότητα που έχουμε να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε ε, και να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Τώρα εκ μέρους ε, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου θέλω να σας ευχαριστήσω και ε, θα σας αναφέρω και, και, που μας δίνετε, και σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία για να έχουμε μια έκθεση σε σχέση με την ευρωπαϊκή πρακτική και πώς θα την αναπτύξουμε. Θέλω να σας παρουσιάσω δύο ομαδοποίησεις ε, των συστάσεων, τις ε, συστάσεις 11 με 16 που έχουν να κάνουν με θέματα ε, διαβαθμισμένων πληροφοριών. Αυτό τονίστηκαν και από τη Συμβουλή για τους και κατόπιν έχουμε τις συστάσεις 16 έως 21 που αναφέρεται σε θεσμικά ζητήματα, δηλαδή μέσω ποιων θεσμών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μπορεί να προβεί στην εποπτεία των οργανισμών ασφαλείας και πληροφοριών. Καταρχήν, ε, το θέμα της πρόσβασης ε, στις απορρίτες πληροφορίες. Η δημόσια πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες ε, αποτελεί ένα θεμελιώδες ε, δικαίωμα που εξυπηρετεί τη δημοκρατική διαδικασία. Παρόλα αυτά, στον τομέα της ασφάλειας και των πληροφοριών υπάρχουν ε, νομίμως κάποιες απόρριτες περιοχές, κάποια απόρριτα στοιχεία και δεν μπορεί το κοινό να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την έκθεση θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει φυσικός, φυσικά διαχωρισμός με μεταξύ τη πρόσβαση του Γενικού Κοινού και των προνόμιων που πρέπει να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με την πρόσβαση που θα έχει σε απόλυτε πληροφορίε ε, στον ε, τομέα τη ασφάλεια και των πληροφοριών. Στη σύσταση 12 λέμε ότι η πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να σχετίζεται με την εντολή υποπτία που έχει και έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν θεσμικοί σύνδεσμοι μεταξύ της πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες και των λειτουργημάτων της υποπτία. Στη σύσταση 13 αναφερόμαστε στο θέμα της διοργανικής ε, συμφωνίας ε, και συστήνουμε ότι πρέπει να υπάρχει διοργανική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, σχετικά με το ΣΥΤΣΕΝ. Αυτό είναι μια ειδική περίπτωση ε, και συμφωνώντα με τον Πρόεδρο δεν νομίζω ότι η σύναψη διοργανικών συμφωνιών είναι μια, μια λύση που πρέπει να ακολουθηθεί γενικά όμως στην περίπτωση ε, του ΣΥΤΣΕΝ φαίνεται να έχουμε ένα μοντέλο λειτουργίας ε, γιατί το Κοινοβούλιο λειτουργεί με ένα τέτοιο τρόπο ε, που προσδίδει και την κατάλληλη θέση στην Επιτροπή Λίμπη να έχει τέτοια πρόσβαση. Σύσταση 14. Εδώ αναφερόμαστε στο ότι πρέπει να υπάρχει ένα γενικό δικαίωμα πρόσβασης ε, ενό επιφορτισμένου οργάνου του Κοινοβουλίου και η ίδια αξιολόγηση ε, θα πρέπει να περιλαμβάνει και το πεδίο αυτή ε, τη πρόσβαση. Επίση, στη σύσταση 15 λέμε ότι θα πρέπει να ε, υπάρχουν συγκεκριμένε κατηγορίε ε, διαφεθυμισμένων πληροφοριών, όπου το Κοινοβούλιο θα έχει πρόσβαση στι πληροφορίε αυτέ χωρί να το ζητάει εκ των προτέρων. Δηλαδή, θα πρέπει να... Ε, του δίνονται, να του δίνεται πρόσβαση σε συγκεκριμένε πληροφορίε, όπω παραδείγματο χάρη στι εξελογήσει απειλών με συγχωρείτε, σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Στη σύσταση 16 ε, εδώ έχουμε λογική ροή, κάτι που προκύπτει από το προηγούμενο και λέμε ότι το όργανο υποπτίας θα πρέπει να είναι το ίδιο που θα έχει και πρόσβαση σε διαβασμένες πληροφορίε. Ε, δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιε θεσμικέ διευθυντήσει, έτσι ώστε να ε, διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που είναι απόρριτες, εξακολουθούν να παραμένουν απόρριτες όταν υπάρχει πρόσβαση του αρμοδίου οργάνου. Εδώ αναφερόμαστε και σε μία λύση όπου το εν λόγω όργανο είναι περιορισμένο σε μέγεθος, έχει περιορισμένο μέγεθος και χρησιμοποιεί διαδικασίες ε, τα ε, ή κάποια μέσα που μπορούν να πείσουν ε, τα ευρωπαϊκά όργανα και τους θεσμούς ότι είναι δυνατό να έχει πρόσβαση το όργανο αυτό σε απορρίτες πληροφορίες χωρίς ε, να παραβιάζεται την απαραίτητη εμπιστευτικότητα για επιχειρήσεις στον τομέα πληροφοριών και ασφάλειας. Σύσταση 18, εδώ αναφερόμαστε στην κατάσταση σε προσωρινή βάση και μιλά υπέρ της Επιτροπής Λίμπη που θα μπορούσε να αναπτύξει κάποιες διαδικασίες τουλάχιστον ε, θα μπορούσε να ξεκινήσει η διαδικασία της εποπτείας και ε, να γίνεται παράλληλα σεβαστός ο χαρακτήρας των απολύτων πληροφοριών. Στη σύσταση 19 είμαστε κατά λύσεων ειδικών επιτροπών Καταρχήν, ε, γιατί δίνουμε, ε, δίνουμε προτεραιότητα ε, στην εποπτεία. Έτσι λοιπόν, καταλήγουμε στην 21η σύσταση και λέμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια Επιτροπή της Λιβύη για την εποπτεία των οργανισμών του χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνη και ασφάλειας. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης εποπτεία και ταυτόχρονα και η λειτουργικότητα των πληροφοριών. Επίσης, ε, ε, αναφερόμαστε και πάλι σε άλλη σύσταση ε, σε, και στο ΣΥΤΣΕΝ που όπως σας είπα είναι μια ειδική περίπτωση και δεν εντάσσεται απαραίτητα στη γενική λύση που προτείνεται στη σύσταση 21. Ολοκληρώνω εδώ, Πρόεδρε, και φυσικά ευχαριστώ να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και όπως είπε και ο κύριος Μπορ, είναι παρόντα και τα υπόλοιπα μέρη τη ομάδα και θα απαντήσουν και αυτέ τι ερωτήσει. Μάλιστα, πολύ ωραία. Τα καταφέρατε, εξαβαστήκατε και το χρόνο και ξεκινούμε τη συζήτηση. Είδαμε ότι ζήτησαν κάποιοι το λόγο. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Ινβελτ. Από ό,τι κατάλαβα, θέλετε το λόγο. yes. Ε, ναι, ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τους παρουσιαστές της μελέτης. Δεν την έχω διαβάσει ολόκληρη γιατί είναι 150 σελίδες αλλά διάβασα μεγάλο μέρος της. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική και ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα γιατί και ως εισηγήτρια για την αξιολόγηση των μέτρων αντιτρομοκρατίας θέλουμε και εμείς να κάνουμε μια παραπομπή εδώ στην παράληψη του θέματος της συνεργασίας των υπηρεσιών πληροφοριών γιατί επειδή αυξάνεται ο αριθμός κακοποιών γενικότερα διαμεθοριακός πρέπει να υπάρχει συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών αλλά με δημοκρατικό έλεγχο. Είχα να πω κάτι σχόλια και ταυτόχρονα ερωτήσεις. Λοιπόν, μία πιο πολιτική. Έχω την εντύπωση από την έκθεση ή μελέτη αυτή ότι η κατανομή μεταξύ ευρωπαϊκής και εθνικής επιτήρησης φαίνεται ότι είναι θέμα θεσμικό, ενώ εγώ νομίζω ότι είναι υποχρέωση που έχουμε προς τους πολίτες, δεν είναι θέμα εθνικών οργανισμών ή ενωσιακών, είναι υποχρέωση που έχουμε προς τους πολίτες. Και άρα όταν λέμε να μην τα πούμε πολύ συγκεκριμένα γιατί μπορεί τότε οι μυστικές υπηρεσίες να έχουν αντιρρήσεις και τα λοιπά. Όχι, δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα. Έχουν και αυτές υποχρέωση προς τους πολίτες και άρα είναι υπόλογες. Επίσης με ενδιαφέρουν όλες οι συστάσεις αλλά ιδιαίτερα θα ήθελα να μιλήσετε περισσότερο για το εξής. Φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη κάποια χάσμα μεταξύ εθνικής και ενωσιακής επιτήρησης γιατί ναι μεν τα οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί δεν έχουν λειτουργικές δικαιοδοσίες αυστηρά αλλά Υπάρχει εδώ μια γκρίζα ζώνη μεταξύ των δραστηριοτήτων εθνικών οργάνων και ευρωπαϊκών τιάφτων, τιούτων μάλλον. Η πραγματικότητα δεν είναι τόσο καθορισμένη όπως λέτε εσείς ως προς τις διαφορετικές δικαιοδοσίες η ευρωπαϊκή επιτήρηση δεν ε, θα αντιγράφει την ε, εθνική, θα τη συμπληρώνει. Δέχομαι τη σύστασή σας να υπάρξει ένα ενιαίο σώμα, αλλά για το Σίτσεν χρόνια μιλάμε, λέτε ότι έχουν τεθεί 7 επισήμως ερωτήματα για το ΣΥΤΣΕΝ νομίζω πολύ περισσότερα είχαν τεθεί. Και έχοντας διαβάσει την έκθεσή σας, βλέπω ότι λέτε ότι ίσως να υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ευρωάστ και Ευρωδίκ, αλλά νομίζω ότι αντί να τονίσουμε κυρίως ελλείψεις των μεν και των δε πρέπει να φροντίσουμε το ΣΥΤΣΕΝ να μπει στη συνθήκη για να ορίζεται εκεί ποιες ακριβώς θα είναι οι ευθύνες του. Δύο τελευταία σχόλια. Κάτι που πρέπει επίσης να εξετάσουμε είναι οι δομές της συνεργασίας μεταξύ μυστικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών πληροφοριών και η σύνδεσή τους με την ιδέα της δημιουργίας ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφορία, πληροφοριών. Τέλος, βλέπω αυτά που λέτε σαν μήνυμα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίξει και αυτό πληρέστερα το ρόλο του, του επιτηρητού και να χρησιμοποιήσει καλύτερα τα υπάρχοντα εργαλεία όποτε θέτουμε ερωτήματα προς το Συμβούλιο και την Κομισιόν, όποτε, δεν παίρνουμε ποτέ ή σχεδόν ποτέ πλήρεις και ικανοποιητικές απαντήσεις. Ευχαριστούμε. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα και σας υπενθυμίζω ότι θα έχει και συνεδρίαση των συντονιστών στο τέλος. Λοιπόν να φροντίζετε όλοι το χρόνο σας. Ο κύριο Κέλλερ. Α, όχι. Λαμπέρτ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι κρίμα που δεν εξετάζουμε ε, την μελέτη για το ΣΕΠΣ μαζί με αυτά διότι και εκεί υπάρχουν ε, συστάσεις οι οποίες όμως διαφέρουν από αυτές οπότε θα ήταν ενδιαφέρον να τα παραβάλουμε διότι Ορισμένα από τα θέματα τα οποία εξετάζουμε δεν αναφέρονται σε κλασικά θέματα ασφαλείας, σε τρομοκρατικές ενέργειες, αλλά είναι και θέματα ε, συνόρων, ε, διαδικασιών. Έχουμε όλα αυτά, όλες αυτές τις οργανώσεις και γι' αυτό θα ήθελα να ε, επανέλθω σε αυτά τα οποία είπε η Σοφή ε, σχετικά με τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα αυτών των οργανισμών. Και ε, από πλευρά εποπτείας <clears throat> πρέπει να εξετάσουμε τι προσπαθούμε να εποπτεύσουμε. Δηλαδή ε, υπάρχουν πολλές φορές όσον αφορά τον, ε, ε, την αναφορά πολλές, πολλά κενά αλλά πώς μπορεί να επανορθωθούν πώς μπορείτε να εντοπίσετε τα κενά και τα λάθη και να τα διορθώσετε μία μελέτη επ' αυτό να πούμε θα ήταν πολύ χρήσιμη Επιπλέον όμως πρέπει να δούμε πώς εσείς ε, ε, μπορείτε να ε, πώς μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις συμφωνίες με τρίτες χώρες γιατί μόνο εάν μπορούμε να εξετάσουμε και αυτό το σημείο υπάρχει κάποιο νόημα στην εποπτεία μας. Επίσης μπορούμε να επηρεάσουμε την, τον καθορισμό του διευθυντή κάποιου οργανισμού διότι πολλές φορές τα διοικητικά συμβούλια εκπροσωπούν εκπροσωπούν απλώς τα κράτη-μέλη, έχουν και ένα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται να έχει κάποιο ρόλο και να μπορεί να παρακολουθεί, να υπάρχει ένας απολογισμός και να βλέπει και τους διευθυντές. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς εσείς αντιλαμβάνεστε αυτή τη διασύνδεση μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πώς θα λειτουργήσει αυτή η συνεργασία, τι μηχανισμός χρειάζεται, διότι ορισμένα κράτη έχουν ε, ήδη πει ότι δεν θέλουν να αναμειχθούμε σε ένα σοβαρό θέμα σαν αυτό. Η κυρία Ρομέρο. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, δεν μπόρεσα να φτάσω νωρίτερα και δεν μπόρεσα να ακούσω τις ε, παρεμβάσεις των προσκεκλημένων για αυτό το πολύ ενδιαφέρον ε, θέμα για τους οργανισμούς ασφαλείας. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με το συντονισμό των, ε, των οργανισμών ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είδαμε πάντα στα φαινόμενα τρομοκρατία, ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν ε, υπάρχει συντονισμό στις πληροφορίες. Το είδαμε όταν είχαμε την επίθεση στι ΗΠΑ όπου οι 16 οργανισμοί πληροφοριών δεν ήταν συντονισμένε μεταξύ τους και το ίδιο συμβαίνει και στην Ευρώπη. Δηλαδή κάθε κράτος μέλο έχει το δικό του οργανισμό, αλλά σε διαφορετικά ε, υπουργεία, σε διαφορετικές επιτροπές, με διαφορετικούς στόχους ε, και παρόλο που έχουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, παρόλα αυτά κάθε χώρα συνεχίζει να έχει τη δική της στρατηγική ασφάλειας με του δικού της στόχου και συνεχίζει ε, να γίνεται πολύ πιο, να καθίσταται πολύ πιο σημαντική η πολιτική της κάθε κυβέρνησης παρά η ευρωπαϊκή στρατηγική. Δεν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός οργανισμός που μπορεί να συντονίσει αυτούς τους οργανισμούς ε, τους εθνικούς οργανισμούς πληροφοριών για να υπάρχει και ανταλλαγή πληροφοριών. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις γίνεται ανταλλαγή των πληροφοριών. Θα ήθελα να ξέρω αν η εποπτεία του Ευρωκοινοβουλίου θα χρησιμεύσει σε κάτι και θα είναι αποτελεσματική, αν πράγματι αυτές οι πληροφορίες δεν ανταλλάσσονται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φυσικά θα ήταν πολύ καλύτερα να κάνουμε τη συζήτηση αν όλοι είχαμε διαβάσει αυτό το έγγραφο. Εγώ ομολογώ ότι δεν το διάβασα μόλις το πήρα τώρα. Αλλά αν κατάλαβα καλά, αυτό το οποίο ε, συζητάμε είναι ότι υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί ασφαλείας και υπάρχει ανάγκη εποπτείας αυτών των οργανισμών. Μάλιστα, αν κατάλαβα καλά, υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί οι οποίοι ήδη εποπτεύουν τους οργανισμούς όπως την Europol, την Eurojust κλπ. Θα ήθελα να ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οργανισμοί αν υπάρχουν, πότε και πώς λογοδοτούν στον Κοινοβούλιο. Δεν έχω ακούσει καμιά φορά να έρθει κάποιος εκπρόσωπος αυτών των οργανισμών εδώ και να μας αναφέρει τι ακριβώς ε, κάνουν και να φέρουν τις εκθέσεις τους στην επιφάνεια. Γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω κάτι για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Herr äh, äh, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω διαβάσει ακόμη ολόκληρη τη μελέτη, αλλά έχω διαβάσει ήδη ορισμένα τμήματα και χαίρομαι διότι τουλάχιστον και εδώ υπάρχει μία ανοιχτή συζήτηση, διότι βεβαίως ε, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες επιτροπές, δεν χρειαζόμαστε νέες επιτροπές, αλλά ε, στην ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα θέλαμε να παραμείνουμε σε ενέργεια σχετικά με την επιτήρηση στα πλαίσια του τρίτου πυλώνα και γι' αυτό έχω και μία ερώτηση προς τα εσάς ιδίω ακριβώς στους οργανισμούς ε, οι οποίοι έχουν εκτελεστικές ε, αρμοδιότητες ε, ή όπου παραπέμπονται όπως παραδείγματος χάρη η Ευρωπόλ όπου μεταφέρουμε τα στοιχεία από τον ένα στον άλλον και διαφορετικά δεν έχουμε καμία συμμετοχή θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένες ισορροπίες συνταγματικές και πάντοτε χρειάζεται να υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος όσον αφορά τα οικονομικά, την οικονομική αυτονομία και την ε, δυνατότητα οργάνωσης. Πρέπει δηλαδή να γνωρίζουμε εάν υπάρχει ένα κοινοβούλιο το οποίο μπορεί να συμμετάσχει στη διαμόρφωση των αρμοδιοτήτων αυτών των οργανισμών διότι ε, άλλο είναι ένα θέμα το οποίο ε, αποφασίζεται απλώς ε, από την περιφέρεια ή από την Επιτροπή και άλλο να συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκπλήσωμε λοιπόν ότι το, η Ευρωπόλ κάνει πάρα πολλές ε, εργασίες σχετικά με την εγκληματικότητα και όχι τόσο πολύ ε, με την οργανωμένη εγκληματικότητα που αναφέρεται σε οχήματα και ε, πρέπει να θα ήθελα να ξέρω πώς αιτιολογείται και πώς διατυπώνεται αυτή η εποπτεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για το έργο σας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το έργο και ιδιαίτερα υπεύθυνη δουλειά σας ε, και τονίζω το θέμα της υπευθυνότητας, ε, γιατί ζητάτε τη διαφάνεια, επιχειρηματολογείτε υπέρ της διαφάνειας και της εχνηλασιμότητας και κάνετε συστάσεις προς αυτή την κατεύθυνση και επίσης δεν ξεχνάτε και την ασφάλεια και την πρακτική εφαρμογή, γιατί και αυτές είναι σημαντικές πτυχές. Μερικές φορές στο Κοινοβούλιο βλέπουμε να υπάρχει αντίφαση μεταξύ των δύο αυτών πτικών ε, εγώ. Έριξα μια γρήγορη ματιά σε αυτή τη μελέτη και παρακολούθησα, μάλλον και είχα και μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με κάποιον από τους συναδέλφους σας ε, πριν κάποιο καιρό. Έτσι λοιπόν, περιμέναμε την προμονησία τη δημοσίευση της μελέτης αυτής. Όπως σας είπα, μπόρεσα να ρίξω μία γρήγορη ματιά, ελπίζω να μην παρεξήγησα κάτι. Θέλω λοιπόν να τονίσω τρία στοιχεία. Η μελέτη τονίζει την πρόταση σχετικά με τη δημιουργία υποεπιτροπής. Ε, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα αυτή. Όμως, εγώ βλέπω τρία προβλήματα εδώ στη σύστασή σας. Ε, λέτε ότι η υποεπιτροπή βασικά θα κάλυπτε τρεις ε, πτυχές. Την ε, πολιτική της διαχείρισης, την ε, πολιτική σκοπιά, τον προπολογισμό, αλλά δεν θα μπορούσε να ελέγξει την επιχειρησιακή πτυχή. Καταλαβαίνω τη λογική σας, πιθανόν να έχετε δίκιο, αλλά να αφήσουμε κατά μέρου τα επιχειρησιακά ζητήματα συνολικά, αν το εκτός από το πεδίο εφαρμογή των δραστηριοτήτων αυτής της Επιτροπής, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να λάβουμε κάποιες σοβαρές αποφάσεις. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση, απλώς ήθελα να επισημάνω ότι αυτό είναι πρόβλημα. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα μεταξύ ΣΥΤΣΕΝ και των υπόλοιπων οργανισμών. Κατανοώ και τη λογική που ακολουθείται εκεί, το ΣΥΤΣΕΝ το κέντρο διαχείριση κρίσεων ε, λογοδοτεί στην Επιτροπή Εξωτερικών Επιθέσεων. Εμεί δεν είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό από οργανωτική σκοπιά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με το θέμα της δημιουργίας της υποεπιτροπής, γιατί στην πραγματική ζωή δεν ακολουθούν τα πάντα τις δικές μας γραφειοκρατικές διευθετήσεις. Μπορώ να αναφέρω, παραδείγματος χάρη, θέματα όπως η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, χρειάζεται για αυτά μια συλλογική προσέγγιση για να αντιμετωπιστούν και να ελεγχθούν. Αλλά νομίζω ότι είναι πρόβλημα αν με συζητούμε για την τρομοκρατία σε μια επιτροπή και για τα υπόλοιπα θέματα σε άλλη επιτροπή, γιατί ε, κάτι τέτοιο θα αφορούσε πολλές αρμοδιότητες από την Επιτροπή. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με τη διαφάνεια. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ορισμένα κράτη-μέλη προφανώς υπάρχουν προβλήματα, αλλά πρέπει να βρούμε μια ισορροπία και να ξεβρούμε την καταλλήλη λύση. Νομίζω ότι το security clearance, αυτή η άδεια των μελών της Επιτροπής είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούν να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο, αλλά θα παραμείνω στα γερμανικά. Ε, ουσιαστικά δεν έχω να προσθέσω τίποτα, έχω όμως μία σύντομη ερώτηση, διότι δεν ξέρω αν αυτό είναι εντός των αρμοδιοτήτων σας, διότι πολλοί από μας εργάζονται στο ψηφιακό τομέα και στην αρχή ε, λέγεται ότι μπορεί κανείς να βρει στο διαδίκτυο αυτή τη μελέτη, αλλά δεν είναι προφανές ε, που μπορούμε να τη βρούμε, σε ποιο ποιο, σε ποια ε, ιστοσελίδα. Θα ήθελα ίσως κάποιες πληροφορίες για να διευκολυθώ στη δουλειά μου. Ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ, η κυρία Κέλλερ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση. Μάλλον ένα σχόλιο και μία ερώτηση. Καταρχήν, το σχόλιο διότι μιλάμε για διαβαθμισμένα έγγραφα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα εμπιστευτικά ε, έγγραφα δεν ε, καθίστανται διαβαθμισμένα ε, εκ του μηδενός, αλλά κάποιος τα έχει κατατάξει σε αυτή την κατηγορία. Οπότε πρέπει να δούμε ποιος τα κατατάσσει και μετά πώς θα τα αντιμετωπίσουμε άπαξ και διαβαθμιστούν. Ε, επίσης, ε, εάν κάνω μία ερώτηση που μπορώ να διαβάσω, τις οποίες μπορώ να διαβάσω να απάντηση στο κείμενο, πέστε μου. Ε, υπάρχει εποπτεία από τα κοινοβούλια για τους συνοριακούς, τους φύλακες των συνόρων και μέχρι ποιο σημείο. Θα ήθελα να μου το διευκρινίσετε και ο κύριος Μπρόντς. Η θέση μου είναι ότι εγώ δεν επίθομαι ε, εύκολα από τα ευρωπα... τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ακόμη λιγότερο για τους μη αμυγός ευρωπαϊκούς. Αλλά υπάρχουν πρέπει να τα παρακολουθούμε και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το κατάλληλο σημείο να διεξαχθεί αυτή η εποπτεία παρόλο που αντιλαμβάνουμε ότι είναι της αρμοδιότητας των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όσον αφορά το θέμα της ε, πρόσβασης των Ευρωβουλευτών στα ε, διαβαθμισμένα έγγραφα θα χρειαζόντουσαν ουσιαστικά περισσότερες διαδικασίες και όχι τόσο μέτρα ασφαλείας, δηλαδή ε, εγώ πιστεύω ότι άπαξ και δεν ε, υπάρχει, ε, άπαξ τα έγγραφα αυτά μπορούν να κυκλοφορήσουν πιο ευρέως, δεν πρέπει να είναι διαβαθμισμένα. Και το ποιος θα έβλεπε τα, τα διαβαθμισμένα έγγραφα έπρεπε ε, να επιλέγεται από, τις, από τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων και άρα από τις πολιτικές ομάδες. Και τίθεται τώρα το ερώτημα ότι οι μη εγγεγραμμένοι δεν, δεν θα έχουν δικαίωμα να πρόσβαση στα έγγραφα αυτά διότι δεν είναι άξιοι εμπιστοσύνης. Ε, και πρέπει να πούμε ότι συμφωνώ ότι δεν πρέπει να είμαστε δεύτερης τάξης πολίτες. Ο κύριος ε, Μπουσουτήλ για ένα τελευταίο θέμα. Ευχαριστώ ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τους συντάκτες αυτής της παρουσίασης. Διάβασα μόνο τις συστάσεις αλλά τις βρίσκω ήδη πολύ ενδιαφέρουσες. Πριν από δύο εβδομάδες ψηφίσαμε, εγκρίναμε τη νέα εντολή του Frontex και πριν ακόμη ακούσω τις συστάσεις σας είχα εκφράσει την ικανοποίησή μου γιατί ζητήθηκαν περισσότερες εγγυήσει για δημοκρατικότερο χαρακτήρα στη λειτουργία αυτού του οργανισμού. Και μετά την ανάγνωση της έκθεσής σας νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση να επωφεληθούμε από τα συμπεράσματά σας για τις επόμενες μεταρρυθμίσεις του. Ένα θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι ακριβώς το θέμα των εμπιστευτικών πληροφοριών. πρέπει, ποια πρέπει να είναι τα όρια του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της πρόσβασης σε εμπιστευτικές πληροφορίες. Ποιες πληροφορίες μπορούν να διατίθενται, ποιες δεν μπορούν να διατίθενται. Τι κανόνες θα μπορούσαν να οριστούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπουσουτήλ. Τώρα οι απαντήσεις. Τους δόκτορες Μπόρν και Σάινεν. Η μελέτη θα διανεμηθεί στα μέλη των εθνικών αντιπροσωπιών που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση που οργανώνουμε την Πέμπτη. Η μελέτη αυτή λοιπόν που μας εξήγησαν, που μας παρουσίασαν οι δύο καλεσμένοι μας. Δόκτορα Μπόρν παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αν μου το επιτρέπετε θα ήθελα πριν απαντήσουμε και οι άλλοι δύο συνάδελφοί μας να... Α, όχι, όχι, εδώ προβλέπουμε άλλη μέθοδο. Εσείς είστε οι καλεσμένοι και αφού ακούσατε τις ερωτήσεις πρέπει να απαντήσετε. Έτσι κάνουμε πάντα. Και επειδή και πάντα καθυστερούμε, καλύτερα να βιαστείτε να απαντήσετε. Καλά. αλλά ήθελα πρώτα να τονίσω ότι συμμετέσχουν κι άλλοι στην ομάδα. Μήπως εσύ Μάρτιν να αρχίσεις πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλα τα σχόλια και ερωτήσεις ήταν ενδιαφέροντα και δεν μπορώ φυσικά να τα απαντήσω όλα, αλλά άκουσα ότι υπάρχει στήριξη για τη δημιουργία υποεπιτροπής σας θα ήταν σωστή μέθοδος νομίζω γιατί θα επέτρεπε το συνδυασμό αποτελεσματικότητας και πρόσβασης σε απόρριτες πληροφορίες για να εφαρμοστεί καλύτερα η εντολή της επιτήρησης. Και έρχομαι έτσι στο ερώτημα του κυρίου Μπουσουτήλ. Δεν μπορεί να προκαθοριστεί νομίζω ποιο ακριβώς είναι το όριο. Ποιες απόρριτες πληροφορίες μπορούν να διατεθούν και ποιες όχι. Η δική μας λύση είναι καλύτερη. Λέμε ότι υπάρχουν κατηγορίες πληροφοριών που μπορούν να χορηγούνται χωρίς προηγούμενη άδεια και υπάρχει και ο καθορισμός από το ίδιο το ενδιαφερόμενο σώμα που καθορίζει μόνο του τι είναι και τι δεν είναι απόρριτο, απόλυτα απόρριτο. Δεν υπάρχει όμως προκαθορισμός. Απ' την άλλη τονίζουμε ότι κάτι ισοδύναμο με τον απόρριτο χαρακτήρα που έχουν οι πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια πάντα θα πρέπει να υπάρχει. Άλλο σχόλιο, αυτά που είπε η κυρία Ρομέρο Λόπες για τον καλύτερο συντονισμό της πληροφόρησης. Αυτό είναι πολύ ακανθόδες πρόβλημα γιατί αν δούμε τρομοκρατικές επιθέσεις ας πούμε μετά κατόπιν εορτής είναι εύκολο να τα συνδυάσει κανείς αλλά αν απλώς έχουμε όλο και περισσότερη πληροφόρηση ασύνδετη που δεν οδηγεί πουθενά δεν έχει νόημα και αυτό και γι' αυτό η προσθήκη όλο και περισσότερων πληροφοριών που έχουν συλλέξει οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν σημαίνει μόνο ότι πρέπει να υπάρξει κατηγοριοποίηση τους αλλά επίσης και κάποια κοινή μεθοδολογία μέθοδοι που να μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε την πληροφόρηση. Αυτό είναι κάτι πολύ πιο απαιτητικό από τον απλό συντονι... από την απλή χορήγηση των πληροφοριών. Γιατί αυτή μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση αντί για μεγαλύτερη πληροφόρηση. Ο δόκτωρ Μπόρν τελευταίος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Έχω κάποια σχόλια, αλλά καταρχήν ε, ε, να σας πω ότι εκτιμώ ότι είχαμε πάρα πολύ πλούσια συζήτηση που, θέτουν ε, τις βάσεις, που θέτει τις βάσεις για μελλοντικές συναντήσεις για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά αν αφήσουμε αυτό κατά μέρος, θα ήθελα να αναφερθώ στα όσα υπόθηκαν σε σχέση με το ότι οι οργανισμοί ασφαλείας ε, ε, δεν θα πρέπει να αποκρύπτουν τι κάνουν από τους οργανισμούς του χώρου ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλειας. Αυτές οι συστάσεις προέρχονται από μια ρεαλιστική σκοπιά. Δηλαδή, εμείς ε, είδαμε ότι αυτοί οι οργανισμοί λειτουργούν σαν το ψάρι στο νερό. Δηλαδή, διαλέγουν ε, την κατάσταση που ε, είναι πιο ευνοϊκή για αυτές. Ε, αλλά αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκέφτεται να δημιουργήσει ένα καλύτερο σύστημα λογοδοσίας, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτή είναι η φύση αυτών των οργανισμών και πρέπει να σκεφτείτε πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό. αλλά νομίζω ότι είναι και δικό μας καθήκον ε, να διασφαλίσουμε ποια θα είναι τα όρια αυτής της εποπτείας. Νομίζω επίσης ότι αναφέρθηκε και το θέμα της έλλειψης συνεργασίας ε, μεταξύ ε, των ε, οργανισμών ασφαλείας και της έλλειψης ανταλλαγής προφορίων. Μπορώ να σας πω ότι αυτός είναι ο σκοπός της εποπτείας, να διασφαλιστεί δηλαδή ότι συνεργάζονται οι οργανισμοί αυτοί μεταξύ τους και Τώρα τα κράτη-μέλη που εξετάζουμε είδαμε ότι τα όργανα εποπτείας εξετάζουν αν σέβονται αυτοί οι οργανισμοί του νόμου, αν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και είναι και αποτελεσματικοί. Έτσι λοιπόν ε, είναι και δικό σας καθήκον ε, να ασχοληθείτε με το θέμα αυτό. Νομίζω ότι θα έπρεπε. Ε, υπήρχε μια ερώτηση για ισορροπία μεταξύ λογοδοσίας και διαφάνειας διαφάνεια. Έχετε απόλυτα δίκιο αλλά νομίζω ότι αυτό που προκύπτει και από τις 22 ε, συστάσεις μας είναι το θέμα της διαφάνειας. Εμείς ε, ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί να δούμε πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με την ε, λογοδοσία και τη διαφάνεια και ίσως κάτι ακόμα. Οι περισσότεροι οργανισμοί ασφαλείας δεν είναι τόσο μυστικοί όσο πιστεύουμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφάνεια και υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που θέλουν ε, να γνωστοποιήσουν. Έτσι λοιπόν ε, δεν σημαίνει ότι μιλάμε για 100% μυστικότητα. Πολλά λαμβάνουν χώρα και στο δημόσιο τομέα. Και επίσης υπήρχε και το θέμα του clearance των μελών του Κοινοβουλίου. Ε, Περισσότερε περιπτώσει. υπάρχει αυτή η άδεια, δίνεται αυτή η άδεια στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να έχουν πρόσβαση ε, σε αυτέ τι ευαίσθητε πληροφορίε, γιατί θεωρείται ότι είναι εκλεγμένοι οι ε, άνθρωποι αυτοί για να επιτελέσουν αυτό το έργο. Θα σταματήσω εδώ, αλλά και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για την ευκαιρία που μας έδωσε για να σας εξηγήσουμε τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τους κυρίους Μπόρν και Σάνιν που μας παρουσίασαν αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα που συζητήσαμε και σας ευχαριστούμε που ήσασταν και συνοπτικοί και σαφιστήκατε το χρόνο. Ωραία, θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Σας ευχαριστούμε. And now, we proceed to point number Kaliningrad. Περνάμε στο σημείο 4 συμπερίληψη της περιοχής του Καλίνιγκραντ ε, στην με παραμαθαρή περιοχή. Θα ακούσουμε εδώ μια παρουσίαση της πρότασης ε, της Κομισιόν για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία του 2006 και κατόπιν. Θα ενημερωθούμε από τον εκπρόσωπο της Πολεωνικής Προεδρίας αν βρίσκεται εδώ και θέλει να πάρει το λόγο και κατόπιν ίσως από τον κύριο Τρενταφυλλίδη που μόλις διορίστηκε εισηγητής για το θέμα του Καλίνιγκραντ. Καταρχήν θα ακούσουμε την Κομισιόν, την κυρία Ζωάννα Τέμπλερ. Είστε εδώ, στην αίθουσα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχω μία πολύ σύντομη παρουσίαση, οπότε θα είναι σύντομη και η πρότασή μου. Ουσιαστικά η διευκόλυνση ε, για την ε, περιοχή του Καλινιγκράτ είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται από καιρού και <clears throat> υπάρχει ε, μία ε, κατάσταση η οποία προβλέπει ότι θα υπάρχουν τρία τμήματα της περιοχής του Καλίνιγκραντ. Το βόρειο μέρος θα μπορεί να κάνει συμφωνία με τη Λιθουανία, το νότιο με την Πολωνία και το κέντρο με την πόλη του Καλίνιγκραντ δεν θα είναι επιλέξιμο. Δηλαδή αυτός ο χώρος θα κατακαιρματιστεί σε τρία τμήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, δημοσιεύσει την δεύτερη έκθεσή της ε, το Φεβρουάριο και ε, επιζητεί συγκεκριμένες λύσεις για τη συγκεκριμένη περίπτωση του Καλίνιγκραντ. Σχετικά με την πολιτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελήφθη πολύ να διατυπωθεί η πρόταση αυτή και όπως βλέπετε και από το κείμενο της ε, ε, προτάσεως κάναμε μια τεχνική, δώσαμε μια τεχνική συνέχεια η οποία ολοκληρώθηκε ε, τέλος Ιουλίου με δύο προϋποθέσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχήν <clears throat> να υπάρχει μία εξαίρεση για τη μοναδική περίπτωση του Καλίνιγκραντ και δεύτερον διότι ο γενικός ορισμός των παραμεθορίων περιοχών λοιπόν όπως προβλέπονται ή στον κανονισμό δεν θα φυγούν και θα δεν θα αμφισβητηθούν. Όταν λοιπόν ε, κοιτάτε το ουσιαστικό άρθρο που είναι το πρώτο άρθρο βλέπετε ότι δεν αλλάζει ορισμό αλλά προτείνουμε να προσθεθεί ένα παράρτημα στον κανονισμό αυτό και ο οποίος θα λέει ότι όλη η περιοχή του Καλίνιγκρατ και ορισμένες περιοχές που διαχειρίζεται η Πολωνία θα θεωρηθούν ε, σαν παραμεθόριες ε, επιλέξιμες περιοχές ε, πέραν αυτών που υπάρχουν σήμερα των 50 χιλιόμετρων. Τώρα, το αν αναρωτιέστε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συμπεριλάβει ε, σαν επιλέξιμες και τις παραμεθόριες πολωνικές ε, περιοχές σαν νέα εδάφη, κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αποδώσει η πρόταση αυτή θα πρέπει να επεκταθεί και στην πολωνική επικράτεια διότι διαφορετικά εάν εφαρμόσετε τον ε, κανόνα των 30-50 χιλιόμετρων ε, οι περιοχές στην Πολωνία θα είναι πολύ μικρές και δεν θα έχουν οικονομικό ή τουριστικό ενδιαφέρον για να υπάρξουν ανταλλαγές. Άρα ε, για να μπορεί να αποδώσει η πρόταση αυτή πρέπει να επεκταθούν τα σύνορα. Επίσης όλες ε, οι διατυπώσεις ασφαλείας ε, που προβλέπει ο παρόν κανονισμός θα συνεχίσουν να ισχύσουν και έχουμε δεσμευτεί να σημειώσουμε τα διευρυμένα σύνορα και να εξετάσουμε την περιοχή αυτή. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. τώρα η Πολωνική Προεδρία, ο κύριος Τζαζίνσκι, μήπως ε, θέλει να αναφερθεί στο θέμα του Καλίνιγκραντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να σας καλωσορίσω όλους ε, εδώ στην αίθουσα, κυρίως στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως βλέπετε δεν πρόκειται για μια τυπική κατάσταση. Ε, η Προεδρία τελικά τυχαίνει να προέρχεται από το, μέλ, από το κράτος μέλος που σε μεγάλο βαθμό θα προέκυπταν ε, πολλά θετικά από την τροποποίηση αυτού του κανονισμού. Για να είμαι σαφής, γι' αυτό μιλώ εκ μέρους της Προεδρίας. Και γι' αυτό σκοπεύω να σας γνωστοποιήσω ήδη ποιο, πώς προχωρούν οι εργασίες στην αρμόδια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και πώς οι συζητήσεις προχωρούν επίσης σε επίπεδο κορεπέρ και Συμβουλίου. Καταρχήν, να παραθέσω το σημείο 4 της παρουσίασης ε, που είδαμε από την πολωνική αντιπροσωπεία στην ομάδα εργασίας για τα σύνορα. Το σημείο 4 αυτής της παρουσίασης PowerPoint που είδαν η όλων των κρατών μελών λέει διαφάνεια έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από τη σκοπιά της πολιτικής αντιπροσωπείας και φυσικά αυτή είναι και η θέση της Προεδρίας. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε από εκεί γιατί αυτό είναι πολύ ζωτικό θέμα. Έτσι λοιπόν αυτό σε μεγάλο βαθμό ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση που ακολουθήσαμε και έναντι των έναντι κρατών μελών. Αυτό που θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε είναι το εξή. Θέλουμε να γνωρίζετε με ακρίβεια ποιες είναι οι τεχνικές διευθετήσεις που θα μπορούσε να δει κάποιος στο μέλλον ε, στην ε, διμερή συμφωνία που υπογράψαμε με τη Ρωσία, η Πολωνία με τη Ρωσία, για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν τρία κύριε ζητήματα που θέλω να τονίσω και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας. Ε, Ευχαρίστω μέσω της γραμματείας της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ να σας γνωστοποιήσω όλες τις ε, λεπτομέρειες ε, των τελευταίων εργασιών μας και τα τρία σημεία που αφορούν την κατέθεση που λαμβάνει τώρα η Πολωνική Αντιπροσωπεία είναι εξή πολιτική χωρίς προηγούμενο. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά να ελέγξουμε αν ένα παρόμοιο σενάριο θα μπορούσε να γίνει κάπου αλλού που δεν έχουμε δει παρόμοια λύση. Έτσι λοιπόν, καθώς αυτή η περίπτωση είναι τόσο συγκεκριμένη, θέλουμε και συγκεκριμένε διθετήσεις. Το δεύτερο σημείο αναφέρθηκε από την Κομισιόν. Και πάλι είναι σύντομο, δεν ε, θέλουμε να αλλάξουμε τον ορισμό. Σε καμία περίπτωση. Σημείο 3. όσα κάναμε πριν ε, δύο χρόνια ε, πριν προσεγγίσουμε την Κομισιόν, υλοποιήσαμε μία ανάλυση κινδύνου και έχουμε σαφή στατιστικά στοιχεία που προέρχονται από αυτή την ανάλυση για το αν θα έχουμε ε, alert σχετικά με το Schengen και δεν ισχύει αυτό. Θα έχουμε τέτοια κατακόρηση. όχι δεν ισχύει αυτό. Και επίσης ε, θα ήθελα να σας πω ότι η Γραμματεία του Συμβουλίου θα παρουσιάσει για κάποιες πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν είναι δυνατό θα υιοθετηθούν δύο δηλώσεις προς αυτό το σκοπό. Η μία δήλωση επιβεβαιώνει και αυτή είναι η διαφεθέτηση με τους Λιθουανούς ότι δεν υπάρχει ε, πολιτική προηγουμένου και η δεύτερη δήλωση εμείς αυτή την ε, ε, δήλωση αυτή η δήλωση είναι της πολεμικής αντιπροσωπείας και εκεί σημειώνουμε όλες τις τεχνικές και πρακτικέ διευθετήσει που θα μπορούσαμε να έχουμε στο μέλλον προκειμένου ε, να διαφυλάξουμε το χώρο Σέγγεν. Δηλαδή, δεν θα έχουμε μια μεγάλη πολιτική, αλλά επαφέ μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των ατόμων. Αυτό είχαμε σκεφτεί από την αρχή και θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Κομισιόν που ρύθμισε αυτή την πρόταση όσο έχει. Είμαι στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και την Πολωνική Προεδρία για την παρουσίαση αυτή. Και τώρα δίνουμε το λόγο στον εισηγητή μας κύριο Τριανταφυλλίδη. Πάρα πολύ σύντομα θέλω να ευχαριστήσω τόσο την Επιτροπή όσο και την Προεδρία για την παρουσίαση αυτής της, αυτού του θέματος. Πιστεύω ότι εκφράζω την Επιτροπή μας, αλλά εν πάση περιπτώσει τη δική μου την ομάδα σίγουρα, καλωσορίζοντας την πρόταση της Επιτροπής ως μια ενέργεια που επιδιώκει να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Προσδοκώ ότι ως Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών δεν θα έχουμε ενδιασμού στην ένταξη του Καλίνιγκρατ στη λίστα των παραμεθόριων περιοχών, καθώς πρόκειται, όπως το υπογράμμισε και η Επιτροπή προηγουμένως, για μια περιοχή που βρίσκεται de facto στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό τον λόγο προβλέπω στη συνεργασία όλων των ομάδων, καθώς και του Συμβουλίου, για την εργασία που ελπίζω θα ολοκληρώσουμε χωρίς ε, αντιδικίες. Επομένως ε, θα καλωσορίσω οποιασδήποτε αντιδράσεις και απόψεις των συναδέλφων ε, και θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση ασφαλώς αφού ακούσουμε και τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Πράγματι σύντομα αυτό θα μας βοηθήσει γιατί Είχαμε προβλέψει 20 λεπτά. Θα δούμε όμως τώρα. κυρία Στάνοκα. Ευχαριστώ ως σκιώδης. Εξ ονόματος των Πρασίνων ήθελα να πω απλώς ότι υποστηρίζουμε την πρόταση. Επειδή και εγώ είμαι εκπρόσωπος της περιοχής εκείνης και εγώ δέχομαι με χαρά αυτή την ιδέα της ελεύθερης κυκλοφορίας και εύχομαι καλή τύχη στην πρόταση αυτή. Ο κύριος Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το ΕΛΚ δεν έχει ακόμα εσωτερικά συζητήσει το θέμα, αλλά από τις σημερινές παρουσιάσεις δεν βλέπω να υπάρξει καμία, κανένα πρόβλημα. Κανείς άλλος, τίποτε άλλο, κανένα σχόλιο. Καμία αντίδραση σε αυτά που μας είπαν ο εισηγητής, η Σκιώδης και ο εκπρόσωπος, ο συντονιστής του ΕΛΚ. Ωραία, περνάμε στο επόμενο σημείο. Εντάξει, στο επόμενο σημείο. Εντάξει, Πολωνική Προεδρία. Ωραία κοινή συζήτηση για τη δέσμη Σένιγκεν, τα σημεία 5 και 6 δηλαδή, για το κεκτημένο του Σέγγεν και τον ε, μηχανισμό αποτίμησης του. Έχουμε τον έμπειρο εισηγητή μας περί τον κύριο Κάρλος Κουέλιο Και θα συζητήσουμε εδώ αυτό το θέμα όπως είπα το κεκτημένο του Σέγγεν και την αποτίμηση των κανόνων λειτουργίας του μαζί με τις τροπολογίες για τον μηχανισμό αποτίμησης της Κομισιόν. Πρώτα λοιπόν η Κομισιόν μετά ο εισηγητής μας κύριος Κοέλιο και μετά συζήτηση. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είναι η κυρία Μπελίντα Πάικ ή η κυρία Μόνικα Μοσχάβερ. Yes, please. Mrs. Belinda Η κυρία Μπελίντα Πάγερ είναι. Α, ναι, χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία μου εδώ. Είμαι υπεύθυνη για τη μετανάστευση στη Γενική Διεύθυνση των Εσωτερικών. Στις 16 Σεπτεμβρίου κατατέθηκε και εγκρίθηκε αυτή η δέσμη που συμπεριλαμβάνει και μία ανακοίνωση καθώς και την αναθεωρημένη πρόταση για το μηχανισμό αποτίμησης και μία τροποποίηση στον κώδικα που ισχύει η λειτουργία του Σέγγεν. Ελπίζω αυτά που μοιράσαμε εδώ να σας ε, βοηθήσουν να καταλάβετε τις προτάσεις αυτές, αλλά να σας κάνω το ιστορικό σύντομα. Το Κοινοβούλιο κατανοεί ότι οι πολίτες θέλουν να απολαμβάνουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας σε ασφαλή εξωτερικά σύνορα. Αυτό είναι ο στόχος λοιπόν, να υπάρξουν ασφαλή σύνορα για να μπορέσει να υπάρξει η ελεύθερη διακίνηση. Έχει έρθει πια ώρα να γίνει η αποτίμηση του μηχανισμού λειτουργίας του Σέγγεν για να δούμε αν μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικός. Αυτό ακριβώς στοχεύουν οι προτάσεις μας. Ο τύπος έχει καλύψει αρκετά αυτές τις προτάσεις αλλά δεν έχει κάνει αρκετή κάλυψη της ανάλυσης που κάναμε για να καταλήξουμε σε αυτές τις προτάσεις. Ήδη στην ανακοίνωσή μας για τη μετανάστευση 4 Μαΐου μαζί με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Ιούνιο και με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούλιο έχουμε καταλήξαμε τελικά σε, αυτά, σε αυτή τη δέσμη που έχει τρία τμήματα. Πρώτον, μηχανισμός αποτίμησης. Δεύτερον, ο κώδικας για τα σύνορα και οι δυνατότητες, οι περιορισμένες δυνατότητες που έχουμε προσωρινά να εφαρμόζουμε ελέγχους στα σύνορα και τρίτον η πολιτική καθοδήγηση που θα μας δώσει κυρίως το Κοινοβούλιο. Πρώτον η αποτίμηση, ο μηχανισμός αποτίμησης. Όπως γνωρίζετε είχαμε ήδη προτείνει τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο ο μηχανισμός αποτίμησης να αλλάξει για να γίνει πιο αποτρεπτικό εργαλείο για να σέβονται τα μέλη καλύτερα τον μηχανισμό αυτόν. Τα προτάσεις εκείνες του περασμένου Οκτωβρίου τις συμπληρώσαμε τώρα και πρέπει να σας πω ότι και κατά την κανονική διαδικασία της συναπόφασης μετά την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου θα συμπληρωθεί επίσης η τωρινή πρόταση. Η τωρινή, το τωρινό νομικό υπόβαθρο είναι το άρθρο 77. Ξέρω ότι τον Ιούλιο το Κοινοβούλιο το τόνισε στη συζήτηση που είχε με την Προεδρία για αυτό το θέμα και το τόνισε επίσης και στο ψήφισμά του τον Ιούλιο. Εμεί συμπεριζόμαστε την άποψή σα ότι το άρθρο 77 είναι η καταλληλότερη νομική βάση για αυτή την πρόταση και γνωρίζουμε επίσης ότι μερικές χώρες μέλη διαφωνούν αλλά συνεχίζουμε να επιμένουμε επί του 77. Τώρα, τα στοιχεία που είναι καινούργια στον μηχανισμό αποτίμησης είναι τα άρθρα 13 και 14. Για να σας βοηθήσω να τα κατανοήσετε και για να δείτε ποια ακριβώς είναι η καινοτομία εδώ τα έχουμε τυπώσει αυτά με πιο παχιά γράμματα. Ό,τι βλέπετε με παχιά γράμματα λοιπόν είναι τα καινούργια στοιχεία. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι να μην υπάρξει μόνο αποτίμηση αλλά και διασφάλιση του ότι αν τα κράτη-μέλη συναντήσουν προβλήματα να μπορούν να την χάνουν κάποιας βοήθειας κάποιο μέλος, χώρα μέλος που έχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και δεν μπορεί επομένως να ανταποκριθεί σε αυτά που προβλέπει το Σέγγεν, τότε να του χορηγείται τεχνική βοήθεια. Αυτή η βοήθεια ελπίζουμε να λύνει το πρόβλημα, αλλά εάν έχουν αποτύχει και όλες οι προσπάθειες υποβοήθησης, τότε να μπορεί η Ένωση να αποφασίζει προσωρινά σε μερικά ή όλα τα κράτη-μέλη να επανέλθουμε στον έλεγχο στα σύνορα για περιορισμένο επαναλαμβάνω χρονικό διάστημα. Τώρα, μετά τη διατύπωση αυτής της πρότασης, τη δυνατότητας δηλαδή προσωρινής επαναφοράς των ελέγχων στα σύνορα, εξετάσαμε τον κώδικα που ισχύει στο Σέγγεν για τα σύνορα. Πρόκειται όπως είπα για έκτακτες και προσωρινές επαναφορές, επιστροφές στους ελέγχους στα σύνορα. Τέτοιες δυνατότητες υπάρχουν για μεμονωμένες χώρες μέλη να επαναφέρουν ελέγχους στα σύνορά τους. Αυτό ήδη αναφέρεται στα άρθρα 23, 24 και 25 του ισχύοντος κώδικα του Σέγγεν. Δεν σκοπεύουμε να αλλάξουμε τη βάση της λήψης αυτών τέτοιων μέτρων. Ο μόνος λόγος για την επαναφορά προσωρινά ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα θα ήταν σοβαρή απειλή στην εσωτερική ασφάλεια μιας χώρας μέλους και αυτή η αποτίμηση πρέπει να μπορεί να γίνεται και εθνικά και ενωσιακά. Δεν είναι σκοπός μας δηλαδή απλώς να διευκολυνθούν να διευκολυνθεί η επαναφορά στους ελέγχους στα σύνορα, αλλά μόνο όταν υπάρχει σοβαρή απειλή και πρέπει να αποδεικνύεται κάθε φορά ότι η προσωρινή αυτή επιστροφή στους ελέγχους θα είναι απαραίτητο μέτρο για την αντιμετώπιση της σοβαρής αυτής απειλής. Αυτό πρέπει να το τονίσω ιδιαίτερα. Επίσης προτείνουμε και νομίζουμε είναι σωστό τώρα που οριμάζει το Σέγγεν η επαναφορά των ελέγχων να απαιτεί λήψη απόφαση σε ενωσιακό επίπεδο. Οποιαδήποτε επιστροφή σε έχει επιπτώσει στη ζωή όλων των πολιτών τη Ένωση. Επομένω, ελέγχους ακόμη και προσωρινά στα εσωτερικά σύνορα έχει επιπτώσεις στη ζωή όλων των πολιτών της Ένωσης. Επομένως η Ένωση έχει συμφέρον να διασφαλίζει τέτοιου είδου αποφάσει να παίρνονται με συνεπή και λογικό τρόπο ενωσιακά. Αλλά τα κράτη-μέλη δεν θα χάσουν τη δυνατότητά τους και μονομερώς να επαναφέρουν τέτοιους ελέγχους αν υπάρχει παραδείγματος χάρη τρομοκρατική επίθεση. Τον Ιούλιο η Σουηδία επανέφερε τους ελέγχους στα σύνορά της για σύντομη περίοδο μετά την σφαγή στη Νορβηγία. Και η Νορβηγία επίσης για, σύντομη, για σύντομο διάστημα επανέφερε τους ελέγχους στα σύνορά της. Όποτε λοιπόν υπάρχουν τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις, μπορεί ένα κράτος μέλος για όχι πάνω από πέντε μέρες και μονομερός να, επιλα... να επαναφέρει τους ελέγχους. Μετά από πέντε μέρες θα χρειάζεται ενωσιακή έγκριση. Τρίτο στοιχείο της δέσμης, πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία του Σέγγεν. Αυτό το αναφέραμε στην σχετική μας ανακοίνωση και θα θέλαμε να προτείνουμε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να κάνουν, μια, να κάνουν τακτικά συζητήσεις κάθε έξι μήνες ας πούμε για τη λειτουργία του Σέγγεν. Ένα είδους υγειονομικού ελέγχου. Εμείς θα σας χορηγούμε την βάση κάνοντας μια εξαμηνία αναθεώρηση του πώς λειτουργεί το Σέγγεν, ποια προβλήματα υπάρχουν και νομίζουμε ότι έτσι θα μπορούσαμε συλλογικά Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Επιτροπή να διαπιστώνουμε ποιες είναι οι εξελίξεις και τι μαθήματα πρέπει να πάρουμε. Έτσι ώστε να μπορούμε και να προβλέπουμε, να αποτρέπουμε προβλήματα, όχι μόνο να αντιδρούμε, αλλά να έχουμε μια πιο συνεπή, πιο μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση για τη διασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας του Σένιγκεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα ας ακούσουμε τον κύριο Κοέλιο, τον συγητή μας. Και κατόπιν θα δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Πολωνικής Προεδρίας και κατόπιν θα ξεκινήσει η συζήτηση. Ο κύριος Κοέλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι συμφωνούμε ότι το σύστημα αξιολόγηση έγκεν που έχουμε σήμερα δεν επαρκεί, είναι ακατόλληλο. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, τουλάχιστον η μεγάλη πλειοψηφία συμφωνεί ότι είναι απαραίτητο και πήγον να καταστήσουμε το σύστημα αυτό πιο απλό και αποτελεσματικό. Αυτό που θέλουμε είναι μια διαφανής εφαρμογή, αποτελεσματική εφαρμογή και συνακτική εφαρμογή του κεκτημένου Σέγγεν. Αυτός ήταν ο στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τότε που μας παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρώτη πρόταση το 2009. Αυτός ο στόχος ε, επίσης αναγνωρίστηκε από το Συμβούλιο ΔΕΗ που έλαβε χώρα το Σεπτέμβριο και το οποίο αναγνώρισε την αναγκαιότητα να ενισχυθεί η εποπτεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τους κανόνες Σέγγεν δίνοντας απάντηση στα ενδεχόμενα κενά και αδυναμίες. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται το στόχο αυτό για μια ακόμη φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή άκουσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ε, την ευχαριστώ των Κομισιόν που απέσυρε την πρόταση που παρουσίασε το 2009 και την αντικατέστησε τον Νοέμβριο του 2010 με νέα πρόταση αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορεί σε συναπόφαση με το Συμβούλιο να μπορεί να δημιουργήσει αυτό το νέο μηχανισμό αξιολόγηση έγκεν. Και επίση ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι δέχτηκε τις περισσότερες από τις προτάσεις ε, που έχουν ε, χορηγηθεί μέσω της δική μου έκθεσης και προσπάθησε να τις ε, θέσει εφαρμογή σε αυτό το νέο πακέτο που μας παρουσίασε. Όπως εξηγήθηκε, η πρώτη πρόταση έχει ως στόχο να τροποποιήσει τη δημιουργία ενός μηχανισμού αξιολόγησης της Σέγγεν και οι μεγάλες αλλαγέ που παρουσιάζονται σήμερα από την Κομισιόν ε, οδεύουν προς την κατεύθυνση αυτή που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε στη δική μου έκθεση είτε στο ψήφισμα που εγκρίναμε στην Ολομέλεια. Δηλαδή, τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ε, πρόσθετη υποστήριξη στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολία και όπου η υπηρεσία Frontex ε, θα πρέπει να έχει έναν ουσιαστικό ρόλο. Και η δυνατότητα ως έσχατη λύση και προσωρινά να μπορεί να υπάρχει νέα εισαγωγή ελέγχων στα σύνορα. Επανεισαγωγή ελέγχων στα σύνορα. Η δεύτερη πρόταση στο τιμό που ευθύναμε στην Κομισιόν ήταν να μας δώσει μια νομική βάση για την εισαγωγή αυτού του μηχανισμού για την πιθανή επανεισαγωγή ελέγχων ε, προβλέπετε στην έκθεση. Χρειαζόταν ε, μια ξεχωριστή νομική βάση, καθώς ε, σημαίνει ότι αλλάζει ο συνοριακός κώδικας έγκεν. Νομίζω ότι με τις προτάσεις αυτές μπορούμε να κάνουμε μια σοβαρή δουλειά και να απρικοδοτήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα πραγματικό μηχανισμό αξιολόγησης έγκεν. Τώρα, είτε από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είτε από την πλευρά του Συμβουλίου. Ελπίζουμε να έχουμε μία κοινή δουλειά, μία αγαστή συνεργασία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, τώρα ε, καλό θα ήταν να ακούσουμε την Πολωνική Προεδρία εάν θέλουν να λάβουν τον ε, λόγο πριν αρχίσουμε τις ερωτήσεις γιατί έχουμε πολλούς οι οποίοι θέλουν να σχολιάσουν και εάν δεν θέλει η Πολωνία να λάβει το λόγο τότε θα έλεγα ότι εφόσον έχουμε πολλούς ενδιαφερόμενους θα πρέπει ο καθένας να μην υπερβεί τα τρία λεπτά για να μπορέσουμε να έχουμε επαρκή χρόνο για καθένα και ξεκινάμε με τον κύριο Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να χαιρετήσω τις προτάσεις αυτές και ε, <clears throat> να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή της καθώς επίσης και τον εισηγητή τον κύριο Κοέλιο. Εγώ είμαι θετικός προς τις προτάσεις αυτές διότι εάν υπάρχει ένα ε, δικαίωμα σαν την ελευθερία διακινήσεως εντός ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν θα πρέπει να, ε, να μπορεί ένα κράτος μονομερός να αφαιρέσει ένα δικαίωμα το οποίο έχει καταρτιστεί πολυμερός και άρα συμφωνώ με την πρόταση αυτή. Αλλά έχω ερωτήσεις όσον αφορά τις πιο πρακτικές διαδικασίες εφαρμογής, δηλαδή πώς θα εξασφαλίσουμε ότι μία απόφαση η οποία λαμβάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι από το κράτος μέλος για την επαναφορά των ε, συνοριακών ελέγχων θα είναι μία απόφαση αρκετά διαφανής και σωστά αιτιολογημένη κατά, τρότον, τρόπον ώστε ε, όλοι να είμαστε ενήμεροι διότι στις αρχές εφέτος οι γαλλικές αρχές είχαν εφαρμόσει ε, ε, συνοριακούς ελέγχους με την Ιταλία για τους γνωστούς λόγους. Αλλά στο νέο αυτό σενάριο με τη νέα αυτή νομοθεσία δεν θα είναι δυνατόν πλέον οι γαλλικές αρχές να κάνουν κάτι τέτοιο μόνες τους. Εντάξει. Τι όμως διασφαλίσεις θα υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να ξέρουμε ότι η απόφαση η οποία έχει ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι ε, σε επίπεδο γαλλικών εθνικών αρχών ε, είναι διάφανο και αιτιολογημένο για να ε, διασφαλίσει και να καθησυχάσει το κράτος μέλος που εμπλέκεται ότι αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες του περί της εθνικής του ασφαλείας και θα μπορούν να υπάρχουν υποκειμενικές αιτίε αντί για αντικειμενικές. Θα ήθελα δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να μας καθησυχάσει επί του θέματος αυτού. Ο κύριος Σενσιού έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι αυτό το νέο νομοθετικό πακέτο που παρουσιάζεται από την Κομισιόν επιφέρει βελτιώσεις ε, στο μηχανισμό Σέγγεν. Δυστυχώς ε, πιστεύω ότι δεν ε, μεταρρυθμίζει πλήρως την διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Φέρου για την ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών. Σε ό,τι αφορά το νέο μηχανισμό αξιολόγησης, είναι πρόταση της Κομισιόν. Έχει συμπεριλάβει κάποιες από τις προτάσεις της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Και η πιο σημαντική είναι το εξής, ότι εισάγεται ένας μηχανισμός ε, κυρώσεων για τα κράτη-μέλη που δεν μπορούσαν να σεβαστούν ε, το χεκτημένο. Το σύστημα αυτό λαμβάνει υπόψη τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Frontex πρέπει να αναλάβουν δράση πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε κύρωσης. Αυτό το σύστημα κυρώσεων μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να ενισχυθούν τα κρατημέλη ε, και να σεβαστούν τα νομικά κριτήρια. Επίσης, ε, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ε, και ενδεχόμενα προβλήματα. Θέλω να τονίσω ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ότι εμείς Υποστηρίζουμε την ιδέα ότι ένα κράτο μέλο δεν μπορεί ποτέ να αποκλειστεί από το χώρο Σέγγεν. Δηλαδή, πάντοτε πρέπει να βρίσκουμε λύσει για να επιλύουμε τα προβλήματα στο πνεύμα τη Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Κάτι ακόμα. Λυπούμαστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανακρίνει ε, την ιδέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υιοθετήσει ένα ενωπημένο σύστημα για τα κράτη-μέλη Σέγγεν και για τις ε, υποψήφιες χώρες καθώς ε, έχουμε, για όσο θα έχουμε δύο διαφορετικά συστήματα αξιολόγησης, θα έχουμε το πρόβλημα των δύο μέτρων και δύο σταθμών. Κάτι που δεσέβεται την αρχή της ίσης Ό,τι αφορά τώρα το μηχανισμό διασφάλισης, η επανεισαγωγή των κατεξαίρεση συνοριακών ελέγχων, των έκτακτων συνοριακών ελέγχων ξεκινά από μία προϋπόθεση που δεν γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης, βάσει της οποίας ότι ε, η προσφυγή σε τέτοιου συνοριακού ελέγχου σε ιστορικό επίπεδο δεν μπορεί να αποτελεί ένα έκτακτο μέτρο. Έτσι λοιπόν η πρόταση της Κομισιόν περιλαμβάνει κάποιες θετικές πτυχές αλλά και κάποιες πτυχές που μας ανησυχούν. Κάτι θετικό είναι ότι ο νέος μηχανισμός απαιτεί οποιαδήποτε απόφαση επανεισαγωγής των συνοριακών ελέγχων θα λαμβάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη σε συγκρίση με το τι ισχύει στο παρελθόν. Όταν ε, κάποια κράτη-μέλη μονομερώς επανσήγαγαν ε, τους συνοριακούς ελέγχους, όπως είδαμε να συμβαίνει στην περίπτωση της Γαλλίας και της Δανίας. Όμως, ε, η δική μας ομάδα θεωρεί ανησυχητικό το ότι η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει ότι οι αποφάσεις αυτές θα λαμβάνονται βάσει επιτροπολογίας. Κάτι που μπορεί να αποκλείσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη συζήτηση. και από τη συμμετοχή στην πραγματική διαδικασία λήψη αποφάσεων. Γνωρίζουμε ότι στη διαδικασία τη επιτροπολογία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πιο περιορισμένο ρόλο. Μια άλλη πτυχή που μα ανησυχεί είναι ότι οι πυλέ ε, κατά τη δημόσια ασφάλεια περιλαμβάνουν και τι μεταναστευτικέ ροέ. Δεν νομίζω ότι οι μεταναστευτικέ ροέ θα πρέπει να αποτελούν λόγο για να επανισάγονται οι έλεγχοι στα ιστορικά σύνορα, θα έπρεπε να έχουμε μία ευρωπαϊκή πολιτική διαχείρισης ε, της μετανάστευσης με ελέγχο στα εξωτερικά σύνορα. Ευχαριστώ. Η κυρία Βέμπερ, αντιλαμβάνομαι ότι όταν το θέμα αυτό πρωτοξεκίνησε στο Κοινοβούλιο, δημιούργησε πολλά ανάμεικτα συναισθήματα, δεν ε, ε, ήρθε λοιπόν μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά μέσω διαφόρων χωρών και χαίρομαι για την αξιολόγηση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον μηχανισμό αξιολογήσεως και ε, χαίρομαι και για τα σχόλια του εισηγητή και του μηχανισμού που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους ε, ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα που προβλέπονται για το μέλλον. Νομίζω ότι η Επιτροπή είναι πολύ σαφής ότι θέλει να περιοριστεί εις ε, τους ε, κινδύνους ε, ασφαλείας και εξωτερικών συνόρων και είμαι σαν να σκέφτομαι μεγαλόφωνα διότι ε, ουσιαστικά εμφανίζει μια ερμηνεία ενώ εδώ μιλάμε για την ουσιαστική νομοθεσία και ίσως καλύτερο θα ήταν να υπάρχει κάποιος ανεξάρτητος όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει τις αποφάσεις και όχι τα κράτη-μέλη με τις ευαισθησίες τους και ε, τις εξάρσεις τους διότι ε, ε, για πέστε μου ποιος ήταν ο κίνδυνος που παρουσιάστηκε ε, στην ε, Ιταλία και πώς αυτό απειλούσε τη Δανία παραδείγματος χάρη. Άρα πιστεύω ότι η κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα θετικό βήμα προς τα ευρώς και, ευρώς και θα μπορέσουμε στο μέλλον να καταλήξουμε σε μία καλύτερη ε, διατύπωση κατά τρόπον ώστε να διασφαλίσουμε όλο το κεκτημένο του Σέγγεν, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό όσο και η οικονομική διακυβέρνηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μάλιστα. Θα ακούσουμε τώρα τους κοιόδης. κυρία Λούτφορντ. Ευχαριστώ, Όπως και οι άλλοι, καλωσορίζω και εγώ τη δέσμη που βασίζεται στην εργασία κυρίως του εισηγητή μας κυρίου Κοέλιο φέτος. Οι δέσμοι είναι πιο λογική, πιο συνεπείς και πιο διαφανής από τις προηγούμενες προτάσεις. Είναι λοιπόν ένα καλό μείγμα στήριξης από τη μία και κυρώσεων από την άλλη. Αυτό νομίζω ακριβώς ζητούσε ο κύριος Κοέλιο και το πέτυχε. Είχα πει για την έκθεση Κοέλιο ότι υποστήριζα μια σύγκληση μεταξύ των δύο συστημάτων αποτίμησης το ένα της λειτουργίας του Σέγγεν και το άλλο των υποψηφίων για το Σέγγεν χωρών και ότι έπρεπε να συμπεριλαμβάνει στοιχεία όπως οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά δωροδοκία. Ελπίζω λοιπόν να εφαρμοστεί η πρόταση αυτή του συγκεκριτή Κάτι άλλο που είχα προτείνει επίσης ήταν η δυνατότητα να μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία να αποτιμηθούν. Όχι ως το δικαίωμα των χωρών αυτών να συμμετέχουν, αλλά και ως δικαίωμα των υπολείπων χωρών να κρίνουν αν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία εφαρμόζουν αυτά που ανέλαβαν. Την δικαστική συνεργασία, την προστασία των δεδομένων κλπ. Δεν είδα τι ακριβώς προβλέπεται για τον τρόπο ακριβώς που θα διασφαλίζεται η συνεργασία αυτή με βάση το άρθρο 77 και τη συμφωνώ ότι είναι η καταλληλότερη νομική βάση αλλά θα ήθελα να πω ότι αν η βάση γινόταν το 70 θα διαφωνούσα το 77 δίνει την απόφαση ενώ το 70 απλή συμμετοχή. Ελπίζω να βρεθεί κάποια λύση και επειδή αναγνωρίζω ότι υπήρξε πρόοδος και ο κύριος Κοέλιο ήθελε μια ρεαλιστική λύση across the channel perspective. This is ελπίζω να γίνει σεβαστό ακριβώς το δικαίωμα των άλλων χωρών μελών του Σέγγεν να αποτιμούν και τη δραστηριότητα της Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεπή εφαρμογή των κανόνων του Σέγγεν είναι ένα άλλο θέμα βέβαια που δεν βασίζεται στην επαναφορά των ελέγχων από τη Γαλλία νωρίτερα φέτος, αλλά και στο θέμα της χορήγησης ημίτων αδειών διαμονής. Η κυρία Στάνο Σκιώδης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Και εμείς χαιρόμαστε για αυτόν τον νέο μηχανισμό και τονίζουμε επίσης ότι για περιπτώσεις που απαιτούν άμεση αντίδραση από μια χώρα μέλος πρέπει να δεχόμαστε έκτακτα μέτρα για τις πέντε μέρες που προβλέπονται. Δεν συμφωνούμε ότι η περίοδος αυτή πρέπει να μπορεί να παραταθεί. Επίσης όπως και οι σοσιαλιστές και σοσιαλίστριες απορρίπτουμε τη σύνδεση μεταξύ μεταναστών και απειλών στη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια έτσι όπως καθορίζεται στο κείμενο. Θα θέλαμε να υπάρχει ένας σαφέστερο ορισμός τι είναι σοβαρή απειλή στην εσωτερική ασφάλεια ενός κράτους. ή σοβαρές ελλείψεις στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Εδώ δεν πρέπει για όλα αυτά να γίνεται παραπομπή στη μετανάστευση επίσης. Δεν μπορούν να επανέρχονται οι έλεγχοι στα σύνορα για περιπτώσεις απλώς επιστροφής μεταναστών. Οι διαδικασίες για όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι σαφείς και πρέπει εδώ το Κοινοβούλιο να τα ξαναδεί όλα αυτά. όταν θα επανεξεταστεί το θέμα της αποτίμησης να παίξει το ρόλο του το Κοινοβούλιο και σε αυτές τις διαδικασίες. Ευχαριστώ. Όχι, εμείς ευχαριστούμε. Η κυρία Κέλλερ τώρα. Βέβαια συμφωνώ με αυτά τα οποία ελέγχθησαν και θα ήθελα να πω ότι παρόλο που συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή, Πολιτική, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ε, διαδικασίες της, στο θέμα αυτό διαφωνούμε διότι η ρητή, ε, η ρητή αναφορά των μετακινήσεων σαν πρόβλημα ασφαλείας ε, δεν με βρίσκουν σύμφωνοι. Δεν συμφωνώ καθόλου μάλιστα. Σχετικά με την κοινοβουλευτική συμμετοχή ακούσαμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά όταν μιλάμε για την απόφαση που πρέπει να ληφθεί για το ποιες χώρες πρέπει να εφαρμόσουν ε, ελέγχου στα σύνορα ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πρέπει να ενημερώνεται για το εάν κάποιος σκοπεύει να κλείσει τα σύνορα και με ποια αιτιολογία. Επίσης ένα άλλο θέμα που μου αφήνει αμφιβολίες είναι τι θα γίνει εάν δεν συμφωνήσει μία χώρα και δεν υπάρχει συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε Στενανταφυλίδης. Είμαι ο shadow rapporteur της ομάδας μου, αλλά μιας και λείπει η κυρία θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την διατήρηση του κεκτημένου του Σέγγεν, μέσω της εισαγωγής ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού αξιολόγησης, ο οποίος δεν θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να εισάγουν μονομερώς, έστω και προσωρινά, ελέγχου στα εσωτερικά του σύνορα. Ωστόσο, η ομάδα μου θέλουμε να τονίσουμε ότι θεωρούμε πως η Επιτροπή δεν άγγιξε το επίδικο στοιχείο του κανονισμού, το οποίο υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει. Τους λόγους δηλαδή σύμφωνα με τους οποίους μπορούν να επαναφερθούν προσωρινά τα εσωτερικά σύνορα των κρατών μελών. Ο κανονισμός ορίζει ότι σοβαρές απειλές στη δημόσια τάξη, στην εθνική ασφάλεια, αποτελούν επαρκείς λόγους για να τεθούν σε εφαρμογή εξαιρέσεις στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται οι ορισμένε συνθήκες που δεν ορίζονται ξεκάθαρα στην νομοθετική πρόταση και η εισρωή ενός μεγάλου αριθμού υπηκών τρίτων χωρών. Το πρόβλημα μιας τέτοιας ρήτρα είναι ότι δεν ορίζονται ούτε οι ειδικέ περιστάσεις, αλλά ούτε και η έννοια της μαζικής εισρωής ανθρώπων. Μπορεί ως πιθανό αποτέλεσμα αυτής της ασάφειας να γίνει κατάχρηση του συστήματος Σέγγεν, καθώς και συγχώνευση των ενιών της μετανάστευσης και του ασύλου. Και τέλος, επιπρόσθετα, έχουμε ορισμένους ενδιασμούς όσον αφορά το ρόλο της Frontex στις περιπτώσεις όπου τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις στην επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων τους, καθώς φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να είναι υποχρεωμένα να δεχτούν αποστολές της Frontex στο έδαφος τους. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ, κύριε Μπρόγκς. Ευχαριστώ. Ο πρόσωπο τη Κομισιόν ε, είπε ότι στην περίπτωση που ένα κράτο μέλος ε, αμελεί διαρκώ τις υποχρεώσει του να ελέγχει τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, θα έχει την αρμοδιότητα να εισαγάγει το δικό τη μηχανισμό συνοριακού ελέγχου χωρί τη συγκατάθεση του κράτου μέλους. Η Κομισιόν δεν μα είπε ποιε εξουσίε θα έχει αν τα κράτη-μέλη. Αν το κράτο μέλο στα εξωτερικά σύνορα είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό στον έλεγχο των εξωτερικών σύνορων. Θα έχει μηχανισμό η Ένωση για να πάρει αντίρρηση παραδείγματο χάρη ε, σε περίπτωση που είναι πάρα πολύ ε, αποτελεσματικό το κράτος μέλος. Φαντάζομαι όχι. Επίσης, ε, και πόσο καιρό δεν μας είπε η Κομισιόν θα έρθουν οι αρμοδιότητες από το κράτος μέλος και θα αναλυφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την η αρμοδιότητα το τελευταίο τελευταία δυνατό εξουσίας η Κομισιόν θέλει να την καταστρέψει αυτή την κυριαρχία του κράτους μέρους. Ε, υπάρχει ένας περιορισμός σε πέντε μέρες ε, και μετά από αυτές η Κομισιόν ε, για άλλους έξι εβδομάδες θα έχει καιρό για να αντιμετωπίσει το θέμα. Και τι θα γίνει εν μεταξύ, θα είναι εντελώς ανοιχτά τα σύνορα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το Ηνωμένο Βασίλειο που προς το παρόν τουλάχιστον είναι εκτός του χώρου Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. σας ακούσουμε την κυρία Ματιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, δεχόμαστε ένα μεγάλο μέρος του τμήματος ε, της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, πολύ θετικά. Φαντάζεστε βέβαια ότι ως ε, Γαλλίδα εγώ θεωρώ ότι το θέμα που αφορά, το τμήμα που αφορά την ε, εισαγωγή των ελέγχων στα σύνορα σε περίπτωση που έχουμε έκτακτες καταστάσεις δεν μου αρμόζει καθόλου και φύγει ένα μεγάλο μέρο τη εθνική κυριαρχία των μελών, των κρατών μελών και δεν νομίζω ότι ο ρόλο τη Κομισιόν ήταν να το προτείνει, ούτε το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο ζήτησαν κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι η Κομισιόν ξεπέρασε τα όρια τη κατά την πρόταση αυτή. Έτσι λοιπόν, μιλάμε εδώ για την επανεσογωγή των συνοριακών ελέγχων σε περίπτωση που έχουμε εκτεκτή ανάγκη. Τι θα γίνει μετά τι πέντε μέρε σε περίπτωση που έχουμε διεξαγωγή των ελέγχων λοιπόν στα σύνορα, πόσο θα διαρκέσει η γνωμοδότηση της Κομισιόν στα πλαίσια της Επιτροπολογίας, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή η γνωμοδότηση θα καθυστερήσει να εκδοθεί και θα ήθελα να μου πείτε πόσο θα διαρκέσει σε περίπτωση που έχουμε εκτεκτή ανάγκη. Και η Κομισιόν μας είπε ε, Παραδείγματο χάρη, αν δούμε μέσα σε πέντε χρόνια πόσε τέτοιε περιπτώσει έλαβαν χώρα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω όμως ορισμένα πρακτικά θέματα σχετικά με την πρόταση και αυτή είναι η δεύτερη πρόταση σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού. Θα ήθελα να ξέρω πώς αυτό θα λειτουργήσει ε, σχετικά <clears throat> με την αλλαγή του κώδικα συνόρων του Σέγγεν του 2006 διότι εδώ βλέπω ότι μιλάμε συγχρόνως και για τεχνικές αλλαγές και υπάρχουν πολλές αλλαγές άρα η πρόταση αυτή θα στηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν ένα κράτος δεν είναι σε θέση να ελέγξει τα σύνορά του, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση. Δηλαδή τι θα συμβεί εάν τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να ελέγξουν τα εξωτερικά του σύνορα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάμψ. Και εγώ ε, θεωρώ ότι η κυρία Γκούντς. Ε, αυτή η ε, πρόταση για την αναθεώρηση των ε, εξωτερικών συνόρων είναι κάτι το οποίο θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Αλλά είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί εδώ επανειλημμένος, διότι το Κοινοβούλιο λέγει ότι είναι απαράδεκτο και ε, θα έπρεπε να θεωρήσουμε ότι για χώρες ε, σαν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία που θέλουν να ε, να ε, συμμετάσχουν στο Σέγγερ ε, ε, θα χρησιμοποιήσουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά ή όλοι θα κρίνονται με τα ίδια μέτρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Βίξτρομ. Όπως είπε ήδη και τόνισε η συνάδελφος κυρία Βέμπερ, εμείς χαιρετίζουμε τη θέση ε, του συγητού και την, ε, το θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το Σέγγεν και είναι ένα θαυμάσιο σύμβολο της ενότητος στην Ευρώπη και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Οπότε στην ε, πρότασή της να τροποποιήσει τον κανονισμό του Σέγγεν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ανέφερε ε, την εισαγωγή συνοριακών ελέγχων στο χώρο του Σέγγεν και αυτό βέβαια πρέπει να τονίσουμε θα πρέπει να είναι μόνο τελευταία λύση απελπισίας και η παράταση των ε, προσωρινών ελέγχων όπως ε, ε, και η άρση του Σέγγεν σε κάποια περιοχή είναι κάτι που θα πρέπει να αποφασίζεται από όλα τα κράτη-μέλη και θεωρώ ότι τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται τώρα είναι απαράδεκτα και δεν μπορούν να παραμείνουν στη διάκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά την εφαρμογή του κεκτημένου του Σέγγεν, συμφωνώ με τις φιλοδοξίες του εισηγητή κυρίου Κοέλιο. Πρέπει να ε, πιστεύουμε στα κράτη αλλά να βασιζόμαστε και στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να το θυμόμαστε. Να μην διακινδυνεύσει σε καμία στιγμή ε, η αρχή της ε, ελεύθερης διακίνησης και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλαμβάνει, να εποπτεύει το σύστημα, να μην αξιολογείται ο κίνδυνος από τα κράτη-μέλη γιατί αυτό διακινδυνεύει την αλληλεγγύη διότι θα έπρεπε ίσως και η Frontex να συμμετέσει στην ανάλυση του κινδύνου για να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θα πρέπει και για τα κράτη-μέλη που είναι ήδη στο Σέγγεν και για τις υπο ψήφιες χώρες να ισχύσουν τα ίδια κριτήρια και ε, να ε, θεωρήσουμε ότι είναι καλύτερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αξιολογήσουμε όλους τους παράγοντες ε, κατά αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ δέχομαι θετικά τις προτάσεις της Κομισιόν, αλλά θα ήθελα να πω ότι κάθε μηχανισμός για να είναι αποτελεσματικός ε, θα πρέπει να έχει σαφείς στόχους, αλλά και παραμέτρους ανάντι και κατάντι και για τους στόχους πιστεύω ότι ο στόχος μας με αυτό το μηχανισμό, στόχος, με αυτό το μηχανισμό Σέγγεν είναι διτός. Να ενισχύσουμε αφενός την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, την εμπιστοσύνη των πολιτών σε ό,τι αφορά την ασφαλειά τους, το ιστορικό των σύνορων Σέγγεν, την εμπιστοσύνη μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών, μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και πρέπει να ενισχύσουμε τη διαφάνεια. Αυτό το θέμα είναι ζωτικό για μένα και το βρίσκουμε και στα τρία σημεία που θέλω να υπογραμμίσω. Καταρχήν, υποδέχομαι θετικά και χαίρομαι που για πρώτη φορά αλλά και για πραγματική φορά εκθέσεις αξιολόγησης θα ακολουθούνται και από συγκεκριμένα μέτρα. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό από την αρχή να έχουμε τα ίδια κριτήρια που θα ισχύουν για όλους και δεν θα υπάρχουν ε, τροποποίησεις των κανόνων του παιχνιδιού και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας να έχουμε αυτή τη διαφάνεια. Αυτή η διαφάνεια θα εξασφαλίσει την ίση μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ε, και δεύτερο σχόλιο για την επανεισαγωγή των ελέγχων πώς ε, θα ε, ορίσουμε μια σοβαρή απειλή και ένα σοβαρό έλλειμμα. Θα προτείνει σαφείς παραμέτρους η Κομισιόν, δηλαδή σε ποιες περιπτώσεις με σαφήνεια μπορεί να αποφασίσει ένα κράτος να επενισάγει τους ελέγχους για τις πέντε ημέρες. Εγώ δέχομαι θετικά αυτή την ιδέα γιατί θεωρούμε ότι αυτό το μετρό θα μας ε, ε, θα επιτρέψει να περιορίσουμε τον πολιτικό χειρισμό αυτού του θέματος ε, και πολλές φορές ε, υπάρχει χειραγώγηση σε επίπεδο εσωτερικό για πολιτικούς λόγους επίσης για τις προτάσεις της Κομισιόν. Δεν θέλει η Κομισιόν να περιορίσει την εθνική κυριαρχία ούτε την ελεύθερη κυκλοφορία. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η πολιτική που ε, ανάγεται σε ένα πιο ευρωπαϊκό επίπεδο θέλει να δημιουργήσει έναν αποτελεσματικό και διαφανή μηχανισμό και έναν επικαιροποιημένο μηχανισμό για να απαντηθούν καλύτεροι οι ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκρουτσέτα. Πιστεύω ότι τι συζητάμε εδώ αυτή τη στιγμή, ότι εμεί ε, μπορούμε να αμφισβητήσουμε και την ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαϊκών πολιτών. Γιατί τελικά, αν έχουμε ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα, ε, θα είναι και για του Ευρωπαίου και για του άλλου. Τώρα, ένα διαφορετικό πράγμα είναι η καταπολέμηση του εγκλήματος. Ε, πολλές φορές μιλάμε και για μεταστευτικές φορές και για έκτακτες καταστάσεις, εκτάκτου ανάγκες. Εγώ νομίζω όμως ότι από τη σκοπιά της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, ουσιαστικά ή γίνεται εδώ, πολλοί θεωρούν ότι πρέπει να οδεύσουμε προς ένα ομοσπονδιακό μοντέλο. Υπάρχει φυσικά και περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών, γιατί η ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών ε, ουσιαστικά ε, σήμαινε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος κυκλοφορία των Ευρωπαϊκών πολιτών και τώρα γίνεται λιγότερο. Επίσης, ε, το θέμα της συνεργασίας των αστυνομιών μεταξύ των κρατών μελών. Ε, αυτό είναι το ζήτημα. Δεν ε, είναι μόνο αποκλειστικό θέμα Σέγγεν, μπορεί να υπάρχουν ε, και πάρα πολλέ απλέ διευθετήσει. Παραδείγματο χάρη, σε διάφορε χώρε ε, μπορεί να έχουν διαπραχθεί ε, κάποια δικήματα και δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο έγγραφο για την απέλαση. Δηλαδή, πρέπει να συμφωνήσουμε για τα μέτρα αυτά. Ότι αν κάποιο ανήκει στο οργανωμένο έγκλημα, δεν μπορεί να βγει από τη χώρα, παραδείγματο χάρη, χωρί να έχει συγκεκριμένα Έγραφα, Γιατί καταπολεμούμε το, τη διακίνηση ναρκωτικών, παραδείγματο χάρη. Ε, το θέμα της μετανάστευσης. Ε, εγώ ειλικρινά πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με αυτά τα τρομερά που συμβαίνουν στη Λαμπεντούσα, εμείς ε, και μαζί μεγάλους βουλευτές, ε, αλλά και σπανούς βουλευτές, υποδεχτήκαμε διάφορους ε, εκπροσώπους που έρχονταν στη Λαμπεντούσα και εγώ πραγματικά δεν είδα εκεί την Ευρώπη που ανησυχεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και για τους δημοκρατικούς θεσμούς γιατί ε, οι άνθρωποι αυτοί στη Λαμπεντούσα αφού τους είχαν πετάξει εκεί για δύο-τρεις μήνες στα ζώα στη Λαμπεντούσα έφτασαν κατόπιν στην Ιταλία, τους έδωσαν ένα ανθρωπιστικό, μια ανθρωπιστική θεώρηση και φτάσανε στα γαλλικά σύνορα και εκεί τους ε, αρνήθηκαν την είσοδο και ε, ξέρετε στο μετών ε, τους έδιωχνε η γαλλική αστυνομία και κοιμούνταν στα δημόσια πάρκα περιμένοντας και στη συνέχεια πέρασαν από τα βουνά. Έτσι λοιπόν το θέμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι είμαστε η Ευρώπη και όταν ε, λέω είμαστε η Ευρώπη, δεν πρέπει να ξεχνάμε όλα τα προβλήματα που έχουμε κατά πολέμηση τη λαθρομετανάστευση. Δεν μπορεί να γίνεται στο χώρο Σέγγεν, πρέπει να γίνεται αλληλέγγυα στα σύνορα της Ευρώπης, στα εξωτερικά σύνορα. Γιατί ε, Όποιο είπε στην περίπτωση αυτή αρνούμε την είσοδο, ε, όποιον έρχεται από την Γαλλία, όποιον έρχεται από την Ιταλία, στην περίπτωση εκείνη ήθελε να απελάσει η Γαλλία ένα την ίσιο παραδείγματος χάρη, δηλαδή τι θα γίνει και εμεί τελικά θα στέλνουμε πίσω στη Μάλτα στου μα έρχονται από τη Μάλτα. Αυτό δεν είναι αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών. Μάλιστα, ο κύριο Κλέη. Ε, ehm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα απλώ να πω ότι η Κομισιόν και οι συνάδελφοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων αλλά αυτό έχει δύο πτυχές ως προς το Σέγγεν τουλάχιστον και το κεκτημένο του. Να, πρώτον να προστατέψουμε τα εξωτερικά μας σύνορα και δεύτερον τις περιπτώσεις όπου κράτη-μέλη δεν μπορούν να διαπράξουν αυτόν τον έλεγχο, να εφαρμόσουν αυτόν τον έλεγχο και τότε θα χρειαστεί τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να αρχίσουν να επανελέγχουν το εσωτερικά του σύνορα λόγω ακριβώς της δυσκολίας αυτής των πρώτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα ήταν δικαιολογημένο να επανεφέρουμε τους ε, ελέγχους στα, σύνορα, στα εσωτερικά σύνορα. Η Κομισιόν λοιπόν προτείνει να αλλάξουν οι ισχύοντες κανόνες μέχρι τώρα και εμείς θεωρούμε ότι οι αρχές αυτές καμιά φορά πρέπει να υπακούν περισσότερο στην πραγματικότητα. Έχω λοιπόν ένα συγκεκριμένο ερώτημα προς την Κομισιόν που έθεσε και ο κύριος Μπρόνς και η κυρία Ματιού. Δηλαδή, αν μια χώρα μέλος για πέντε μέρες επαναφέρει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, και αυτό δημιουργήσει ολόκληρη διαδικασία συζήτηση επιτροπολογίας για παράταση των μέτρων σε αυτή την περίπτωση τότε η Κομισιόν θα εξετάζει το θέμα για έξι εβδομάδες και μετά θα γίνεται μια αποτίμηση, αξιολόγηση και μετά ξανά προτάσεις και αυτό μπορεί να κρατήσει τρεις μήνες. Τι θα κάνουμε όμως αν η κατάσταση είναι επίγουσα μετά τις πέντε, πέντε πρώτες μέρες. Ποια διαδικασία ακολουθείτε. Και όσο περιμένει η χώρα μέλος την έγκριση της παράτασης, τι θα γίνει όσο περιμένει. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Λόπες. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι ότι οτιδήποτε σοβαρό συμβαίνει στην Ευρώπη μπορεί να θεωρηθεί σαν σοβαρή απειλή στην εσωτερική τάξη ενός κράτους μέλους. Ούτε μιλάμε για τεράστιους αριθμούς εγκληματιών που θα απειλήσουν την Ευρώπη. Μιλάμε για εξωτερι... εξαιρετικές περιπτώσεις παραδείγματο χάρη αυτά που δημιούργησε η κατάσταση στη Λιβύη και που οδήγησαν στην επαναφορά ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα το να λέμε ότι αυτά είναι απειλή στη δημόσια τάξη, εσωτερική δημόσια τάξη θα ήταν το ίδιο σαν να λέγαμε ότι όποιος ζητάει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εγκληματίας ή συνεργάζεται με δουλεμπόρους. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τέτοιου είδους φιλοσοφία να συζητιέται γιατί η ανασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν οφείλεται κυρίως στην πλημελή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ασφαλείας στο σύνολό του. Και αυτό με τη σειρά του οφείλεται στο ότι επί πολλά χρόνια η Ευρώπη δεν είχε κανένα μηχανισμό ασύλου. Μέχρι να υπάρξει κάποιος μηχανισμός να λυθεί αυτό το πρόβλημα, τότε όλο αυτό τον καιρό που θα λείπει η Ευρώπη θα αντιμετωπίζει όντως προβλήματα που θα δικαιολογούν όλο και περισσότερη επαναφορά στους ελέγχους. Γιατί η συνεργασία με γειτονικέ μας χώρες είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό, για ιδίως γύρω από τη Μεσόγειο. Και το μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι υπέρ της δημοκρατίας στην Αλγερία, τη δημοκρατία, στην Αλγερία, την Τινησία, το Μαρόκο, τη Λιβύη όταν θέλουμε να δώσουμε αυτό το μήνυμα, δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να λέμε ότι θα έχουμε όλο και περισσότερους εσωτερικούς ελέγχους γιατί υπάρχουν σοβαρές απειλές στη δημόσια τάξη. Γιατί αυτό θα σήμαινε ότι λέμε κάτι γελίο στην ουσία, κάτι προσβλητικό. Δεν έχει καμία σχέση με ευρωπαϊκές αξίες και μου φαίνεται ότι είναι κάτι σκανδαλώδες. Και Μιλάμε για την εθνική κυριαρχία, μιλάμε για το έγκλημα. Όταν φυσικά έχουμε μια τρομοκρατική επίθεση στην Ορβηγία, είναι ένας λόγος. Ε, ξαφνικά η στρατηγική που έχει η Ευρώπη για τη στρατηγική να τεθεί σε εφαρμογή. Όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με το τι συνέβη στη Μεσόγειο. Δεν έχει καμία σχέση με το τι συνέβη λοιπόν στη Μεσόγειο. Έτσι λοιπόν αυτό το μέτρο προτείνει η Κομισιόν. Δεν θα ήταν κάτι απαραίτητο αν τα κράτη-μέλη είχαν διαχειριστεί καλύτερα και είχαν ε, τους ε, αρμόδιους πολιτικούς ε, για να χειριστούν καλύτερα αυτές τις κρίσεις. Υπάρχουν επαρκείς οδηγίες που αν είχαν τεθεί σε εφαρμογή τότε δεν θα χρειαζόταν αυτός ο μηχανισμός που παρουσιάζεται σήμερα εδώ και είναι πολύ κακό μήνυμα αυτό για τη συνεργασία στη Μεσόγειο. Αυτό ήταν το επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε θα ήθελα να ακούσω εδώ την εκπρόσωπο ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτού δώσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Κοέλιο. Ευχαριστώ. Θα κάνω ορισμένες παρατηρήσεις και θα δώσω λόγο και στον συνεργάτη μου κύριο Μόσχαμερ ε, σχετικά με το πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα αυτό για να δούμε πώς ε, θα αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις εκτά του ανάγκης που υποχρώνουν τις χώρες να ε, επαναφέρουν τους συνοριακούς ελέγχους. Εμείς δεν θέλουμε νέα βάση ε, για την εφαρμογή συνοριακών ελέγχων ε, και ε, μόνο θα επιτρέπονται εάν υπάρχει σοβαρή, σοβαρός κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Δηλαδή πλούστατα συμφέροντα μειονοτήτων δεν επαρκούν αντιθέτως στον κώδικα Schengen δεν προβλέπεται ότι η αξιολόγηση των κρατών μελών θα πρέπει να αποδείξει ότι η εισαγωγή προσωρινά των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων είναι αναγκαστικό αλλά και λογικό μέτρο. Δεν πρέπει μόνο να αποδείξουν ότι υπάρχει σοβαρή απειλή για την δημόσια ασφάλεια αλλά θα πρέπει συγχρόνως να ε, υπάρξει μία απόδειξη ότι δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για την αντιμετώπιση χωρών που δεν είναι στο Σέγγεν σε σχέση με αυτόν που ήδη είναι μέλη. Το κεκτημένο του Σέγγεν όμως ε, ισχύει για τις χώρες Σέγγεν και για τις χώρες οι οποίες επιθυμούν να προσχωρήσουν στο σύστημα αυτό. Ε, κάποιος ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στις κατευθυντήριες ε, ε, γραμμές σχετικά με τις επικοινωνίες, τα ταξιδιωτικά έγγραφα κτλ. Έχουμε συζητήσει τα θέματα αυτά με ορισμένα κράτη-μέλη, διότι οι κατευθυντήριες γραμμές που στηρίζουν την εφαρμογή του κεκτημένου του Σέγγεν πρέπει να εφαρμόζονται και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή μέχρι το τέλος τέλος του έτους. Προτού λοιπόν ε, περάσω το λόγο στον ε, συνάδελφό μου, θα ήθελα να σας πω ότι εδώ δεν υπάρχει αντιπαράθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με, ε, το, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν προσπαθούμε να προκαταλάβουμε τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία είναι υπεύθυνα για το τι ε, γίνεται στις χώρες τους αλλά η εμπλοκή μας στα εξωτερικά σύνορα ε, είναι τριολογημένη και ε, δεν προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε τους δικούς μας ελέγχους στους συνήθεις ελέγχους της αστυνομίας. Ο συνάδελφός μου θα σας πει πώς λειτουργεί η διαδικασία και του δίνω το λόγο. Κύριε Μοσχάμερ, εξ ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα σας παρακαλώ αν έχετε διευκρινήσεις, κυρία Μοσχάμερ, να τις παρουσιάσετε. Κοιτάξτε, θα παρουσιάσω πολύ σύντομα ε, όσα ακουστηκαν. Έχουμε δύο διαδικασίες, διαδικασία εξέτασης που θα ισχύει για περιπτώσεις που προβλέπονται για την επανεισαγωγή των ε, συνοριακών ελέγχων. Ε, εδώ μιλάμε περίπτωση χάρη όταν έχουμε κάποιες αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις. Στην περίπτωση αυτή το σχέδιο μέτρου θα υποβαλόταν στην Επιτροπή Κομίτη και θα ενημερώταν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί ε, έχουμε τα εκτελεστικά μέτρα όπως το έχουμε στο κανονισμό. Ε, το 22 πρέπει να ενημερώνεται το Συμβουλίο και το Κοινοβούλιο ταυτόχρονα. Η Κομισιόν μπορεί να προχωρήσει μόνο αν υπάρχει ειδική πλειοψηφία για να γίνει κάτι τέτοιο. Αν υπάρχει ειδική πλειοψηφία να μην προχωρήσουμε, τότε η Κομισιόν δεν μπορεί να θετήσει τη διαδικασία. Δεν μπορεί να θετήσει το μέτρο σε ό,τι αφορά τώρα την διαδικασία έκτακτη ανάγκη. Μετά από πέντε μέρε η Κομισιόν μέσα σε κάποιε ώρε θα είναι σε θέση να υιοθετήσει την απόφαση. Δεν μιλάμε για έξι εβδομάδε. Μέσα σε λίγε ώρε η Κομισιόν θα ήταν σε θέση να αποφασίσει για την παράταση ε, του συνοριακού ελέγχου. Αυτό το μέτρο θα υποβαλλόταν στην Επιτροπή Κομίτη και αν διαφωνήσει η Επιτροπή τότε δεν μπορεί να εφαρμοστεί η απόφαση περαιτέρω για την, τον αριθμό των περιπτώσεων που είχαμε από τότε που υιοθετήθηκε ο συνοριακό κώδικα, Μιλάμε για 26 περιπτώσει. Ε, τι αναλύσαμε λεπτομερώς και αυτό μα οδήγησε στι 5 ημέρε, για τι ε, οποίε μπορούν ε, να επανεισάγουν του συνοριακού έλεγχου στα κράτη-μέλη αν χρειάζεται άμεση δράση γιατί σε καμία από αυτέ τι περιπτώσει ε, κανένας έλεγχο δεν διήρκησε περισσότερο από 5 μέρε. Γι' αυτό η Κομισιόν πρότεινε τις πέντε μέρες. Πιστέψαμε ότι ήταν ε, ο επαρκής χρόνος με τη δυνατότητα παράτασης αν χρειαστεί. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Σας ξαναδώσουμε το λόγο στον κύριο Κοέλιο. Ευχαριστώ. Θα είμαι σαφής. Οι προτάσεις της Κομισιόν οδεύουν προς την κατεύθυνση. Ευχαριστώ την Κομισιόν για την πρωτοβουλία αλλά φυσικά πρέπει να εργαστούμε περιορισμένων λεπτομεριών. Θέλω να υπογραμμίσω όσα είπαν οι συνάδελφοί μου σχετικά με τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Νομίζω ότι και ευχαριστώ την Κομισιόν την απάντηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πιο σαφέ αυτό το θέμα στα έγγραφα, ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για υποψήφιε χώρε και κράτη που είναι ήδη μέλη του χώρου Σέγγεν. Λοιπόν, να σας πω τι προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να έχουμε ένα σύστημα αξιολόγησης που να λειτουργεί. Γιατί πολλοί ομιλητέ είπαν και ορθώς ότι ο ομότιμος έλεγχος δεν λειτουργήσε. Δεν λειτουργήσε. Γιατί κάθε κράτο μέλο κάνει ένα παζάρεμα, μια ανταλλαγή για να μην υποχρεωθεί να ακολουθήσει τους κανόνες 100%. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε ένα κοινοτικό σύστημα με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη συμμετοχή της υπηρεσίας μας, του οργανισμού Frontex, προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα. Αλλά αν θέλουμε το σύστημα να λειτουργήσει θα πρέπει να απαντήσουμε και στο ξεσερώτημα. Τι θα κάνουμε όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα σε ένα κράτος μέλος. Τώρα, αυτή τη στιγμή αν έχουμε αξιολόγηση ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε εξωτερικό σύνορο, τίποτα δεν συμβαίνει. Δεν υπάρχει κανένα εργαλείο, κανένα μέσο για να αναγκαστεί το κράτος μόλις να αντιδράσει. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξεβρούμε ένα σύστημα προκειμένου τον λόγο κράτος μέλος, αν ε, λάβει ενημέρωση που θα λέει ότι ο έλεγχος που διεξάγεται στα εξωτερικά σας σύνορα δεν λειτουργεί, θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και να ξαναπώ, η πρώτη αντίδραση θα πρέπει να είναι μία προσέγγιση κοινή. Δηλαδή η Frontex, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσουν το κράτος μέλος να επιλύσει το πρόβλημα, αλλά αυτό θα πρέπει να το <laughs> δούμε και να δούμε τι θα κάνουμε αν παραμείνει το πρόβλημα. Γιατί τότε θα έχουμε πρόβλημα ασφαλείας, όχι μόνο σε εκείνη τη χώρα, αλλά σε όλες τις χώρες. Γιατί μία δυναμία στον έλεγχο εξωτερικού συνόρου σε μία χώρα αποτελεί πρόβλημα ασφαλείας για όλο το χώρο Σέγγεν. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη επανοσεγωγής των συνοριακών ελέγχων. Και όπως ε, πολύ καλά είπε ο κύριος Σέντσιου, θα πρέπει να μιλάμε για ένα έκτακτο και προσωρινό μέτρο. Μόνο για το χρόνο που χρειάζεται, προκειμένου να επιληθεί το πρόβλημα. Και συμφωνώ με τον κύριο Έντσιου και στο εξή. Έχω και εγώ αμφιβολίε αν η επιτροπολογία είναι ο καλύτερο τρόπο να τα αποφάσει για τα θέματα αυτά. Το δικό μας όμως πρόβλημα, κατά την άποψή μου, θα είναι ε, σχετικά με το ζήτημα που ανέφερε ο κύριος Μπουζουτήλ. Είπε, πηγαίνουμε ως ένωση ως Ένωση συντεταγμένα θα αντιμετωπίσουμε την ε, απειλή που μπορεί να προκύψει για την ιστορική ασφάλεια ενός κράτους μέλους. Νομίζω ότι εδώ έγκυται το πρόβλημα. Και θα πρέπει σοβαρά να το σκεφτούμε αυτό. Θα πω τρία πράγματα σχετικά. Καταρχήν, δεν γνωρίζω αν θα πρέπει να ακολουθήσουμε το βήμα αυτό. Δηλαδή, αν θα έπρεπε να δεκτούμε η κοινότητα ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, δηλαδή σε ένα κρατό μέλο. Γιατί όπω η Κομισιόν μα είπε, η αρμοδιότητα για την ε, εσωτερική δημόσια τάξη είναι αρμοδιότητα του κάθε κράτου μέλου, τη κάθε κυβέρνηση. Δεύτερον. Τώρα, κάθε κράτο μέλο έχει το δικαίωμα να επενδύσει για του συνοριακού ελέγχου για 30 ημέρε με δυνατότητα παράτασης όσες φορές θέλει. Είναι λογικό να σκεφτόμαστε ότι το Συμβούλιο θα δεχτεί μείωση σε πέντε ημέρες και πάνω από τις πέντε ημέρες θα πρέπει να ζητήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύουμε ότι το Συμβούλιο θα δεχτεί κάτι τέτοιο. θέλουμε να ενδυναμώσουμε το μηχανισμό αξιολόγηση έγκαι. Νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μια ενωσιακή προσέγγιση, αλλά θα πρέπει να επιζητήσουμε και μια λύση που να μπορεί να εγκριθεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε στο Συμβούλιο. Αν τελικά έχουμε πάρα πολλέ ε, πολύ κάθετη στάση και ενδυνεύουμε τελικά να χάσουμε τα πάντα. Πρέπει να ενισχύσουμε το χώρο Σέγγεν με κάποιες λύσεις. Κάποιος υπερθύμισε την Ορβηγία. Αναφέρθηκε στο τι συνέβη στην Ορβηγία. Αυτό είναι καλό παράδειγμα. Στην Ορβηγία η κυβέρνηση με για τους συνορικούς ελέγχους για δύο ημέρες από όσο θυμάμαι, για 48 ώρες. Γιατί δεν ήξεραν τι συμβαίνει. Δεν ε, ήξερα αν πρόκειτο για ένα μονομένο δολοφόνο ή για εγκληματικό δίκτυο, δίκτυο εγκληματιών, συμμορία. Έτσι λοιπόν ε, αποφάσισαν ε, να, έχουν, να επανεισάγουν τους ελέγχους, όλοι συμφώνησαν, κατόπιν συνειδητοποίησαν ότι πρόκειτο για ένα και μόνο άτομο και κατήργησαν το συνοριακό έλεγχο. Αλλά τι θα συνέβαινε αν δεν μπορούσαν να βρουν τον άνθρωπο αυτό επί τόπου και πολύ γρήγορα ή αν δεν μπορούσαν να έχουν επαρκείς αποδείξεις για να αξιολογήσουν ότι δεν πρόκειται για δίκτυο εγκληματικό. Αν χρειαζόταν δηλαδή μία-δύο εβδομάδες, ένας μήνας. Και θα έπρεπε να έχουν ε, του ελέγχου στα σύνορα. Με αυτό το σύστημα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να ζητήσουν την άδεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν η απόφαση μπορούσε να ληφθεί από το Συμβούλιο, γιατί η Νορβηγία δεν είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα επιτρεπόταν να λάβει μια απόφαση για τα εσωτερικά σύνορα στη δική του έκταση, στη δική του επικράτεια. Δηλαδή μιλάμε για διαφορετικές καταστάσεις που πρέπει να εξετάσουμε πολύ σοβαρά. Κύριε Πρόεδρε, τα λέω μα. Χρειαζόμαστε μια κοινωτική προσέγγιση για το σύστημα αυτό. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να αξιολογεί ουδέτερα το κάθε κρατό μέλο. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα όπου οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και κυρίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υποστήριξη τη Frontex και την υποστήριξη του Κοινοβουλίου μπορούν να υποχρεώσουν τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν τους κανόνες Σέγγεν, να ακολουθήσουν του κανόνε Σέγγεν, αλλά πρέπει να εγκρίνουμε τι λύσει αυτέ. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να διατηρήσουμε μια ισορροπία. Ελπίζω στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πετύχουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κόλλιο. Έχουμε καθυστερήσει ως συνήθως. Και θα πρέπει... Λοιπόν να θυμόμαστε ότι έχουμε περιορισμούς και βλέπω ότι ορισμένοι δεν συμφώνησαν με τη σκέψη και τη συλλογιστική του κυρίου Κοέλιο και ότι η κυρία Μπότσκουρτ ε, ε, δεν συμφωνούσε αλλά από ό,τι ξέρω ο εισηγητής έχει τον τελευταίο λόγο σε μια συζήτηση. Εάν θέλετε κάτι να πείτε έχετε 30 δευτερόλεπτα για να μπορέσει να δευτερολογήσει ο κύριος Κοέλιο γιατί νόμιζα ότι σηκώσετε το χέρι σας γιατί κάτι θέλατε να συζητήσετε την ώρα που παρουσίαζε τη συλλογιστική του. Όχι, δεν θα να κάνω ερώτηση στον κύριο Κοέλιο, απλούστατα δεν μου απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό που ρώτησα και γι' αυτό επανήλθα. Εντάξει, τότε αν ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας προτείνω να χρησιμοποιήσετε τη γραπτή διαδικασία για να πάρετε περαιτέρω διευκρινήσεις. Υπάρχει πάντα αυτή η δυνατότητα, αλλά γιατί είμαι εδώ τότε εδώ ή ακούω, κάνω ερωτήσεις, γιατί ποιος είναι ο λόγος να παρίσταμε αν πρόκειται να ε, έχω γραπτή απάντηση. Θέλετε να απαντήσετε αν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί πολύ σύντομα να σας απαντήσει. Η ερώτησή μου... ότι εκτός από τη νέα πρόταση Υπάρχει και η τροποποίηση ε, ε, των ελέγχων ε, των σειρώνων σύμφωνα με το Σέγγεν και την απόφαση του 2006. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν πρόκειται να υπάρξει μία αλλαγή σχετικά με τον συνοριακό κώδικα του 2006 και το άλλο θέμα ήταν σχετικό με τις ε, τεχνικές αλλαγές. Αλλά εφόσον αλλάζει τα συμφραζόμενα στο ένα θέμα, ίσως αλλάζουν και σε άλλα σημεία. Και επίσης πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη δεν θα προφασιστούν ε, ε, αδυναμία για να μην καλύπτουν τα σύνορά τους όταν έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν εις τους συνοριακούς ελέγχους. Κυρία Χολμάγερ, με συγχωρείτε η κυρία Μόσχαμερ μπορεί να απαντήσει σύντομα. Ευχαριστώ. Ε, ερχόμαστε περίπου από την ίδια περιοχή αλλά δεν υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των προτάσεων τις οποίες ε, προ, ε, ε, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των τροπολογιών του, 2000, του Μαρτίου 2011. Ε, διότι σύμφωνα με τον κώδικα του 2006 και όπως ε, εφαρμόζεται ε, έχει ήδη υποστεί αλλαγές σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Άρα η πρόταση του Μαρτίου ισχύει τώρα και δεν υπάρχουν επικαλύψεις. Όσον αφορά την ερώτησή σας για το πώς θα διασφαλίσουμε ότι ε, θα μπορέσει να υπάρχει ε, έλεγχο των εξωτερικών συνόρων από τα κράτη-μέλη, τα κράτη είναι υποχρεωμένα. Ε, στηρίζονται και οικονομικά και τεχνικά για αυτό το λόγο και οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα και η άρση είναι τελευταία λύσεις ε, ε, ευχαριστώ για την συντομία της κυρίας Μοσχάμερ και τώρα θα μας μιλήσει ο κύριος Κάσμαν σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Είχαμε μία πρόταση το 2008, τροπολογίες το 2009, μετά ίση στη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, δεύτερη έκδοση του σχεδίου εκθέσεως από τον κύριο Κάσμαν, τον εισηγητή που θα παρουσιάσει την πρότασή του και ε, θα θα μπορέσουν ε, να, να υποβληθούν τροπολογίες μέχρι 10 Οκτωβρίου σε μια εβδομάδα δηλαδή, δεν είναι πολύ χρόνος και η ψηφοφορία θα γίνει τον ε, Νοέμβριο. Κύριε Κάσμαν έχετε το λόγο. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε μου λέτε πόσο χρόνο έχω. Είχαμε προβλέψει μισή ώρα αλλά δεν είναι το τελευταίο θέμα που είχαμε πριν τη συνεδρίαση των συντονιστών. Οπότε όσο, όσο πιο σύντομος είσαστε τόσο καλύτερα. Θα είμαι εξίσου σύντομος με την απάντησή σας η ιστορία αυτή όπως είπατε ανέρχεται στο 2008 και εντωμεταξύ ε, υπήρξε μία ε, καθυστέρηση ε, της ψηφοφορίας μετά την πρώτη ανάγνωση διότι επανήλθε στην συνομοθετική διαδικασία το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ δεν έχει υποβάλει τροποποιημένη πρόταση. Η πρωτοβουλία είναι στα χέρια του Συμβουλίου και μάλλον ε, το, ε, το Μάιο η Επιτροπή ε, υπέβαλε μια δεύτερη πρόταση οπότε έκθοτε η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων αποφάσισε να συγχωνεύσει τη δεύτερη πρόταση με την πρώτη και με αυτόν τον τρόπο να καταρτήσει μια νέα έκθεση, πράγμα το οποίο έκανα. Εν τω μεταξύ, ο Επιτροπής Σεύκοβιτς έγραψε στην διάσκεψη των Προέδρων και είχε την ευγένεια να μου στείλει ένα αντίγραφο και ε, διατυπώνει τις ανησυχίες του ότι αλλάζουμε ε, τον κανονισμό 1049 κατά αυτόν τον τρόπο και ε, συγχωνεύουμε τις δύο προτάσεις. Ενώ αυτός πιστεύει ότι θα έπρεπε να ασχοληθούμε μόνο με την πρόταση της Λισαβόνας, τη δεύτερη πρόταση, και μετά να γίνει αργότερα μία γενική ανάταξη του κειμένου αλλά θεωρήσαμε ότι δεν ήταν σωστό αυτό και θα ήταν και αδικαιολόγητο. Πώς θα εξηγήσουμε στους πολίτες ότι δεν χρησιμοποιήσαμε τη μόνη πολιτική ευκαιρία που είχαμε να αλλάξουμε τον κανονισμό 1049 του 2001 κατόπιν των ψηφισμάτων που ανέρχονται στο 2006 και ιδίως κατόπιν των εκθέσεων Σαργεντίνη και Χάουταλα που είχαν υπερψηφιστεί πανηγυρικά το Σεπτέμβριο. Ε, οπότε γι' αυτό τα θέματα τα οποία εξετάσαμε, η εξέταση Επιτροπή και εμείς, ήταν ε, το άρθρο 15 υποπαράγραφος 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας που πρέπει να περιλαμβάνεται στον κανονισμό για να μπορεί να ισχύσει σε σχέση με τους οργανισμούς και τις επιτροπές που καταρτίζονται από το θεσμικό από τα θεσμικά αυτά όργανα, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τη Frontex κτλ. Κατόπιν αυτού ε, ζητήσαμε να έχουμε μια ε, νομική γνωμοδότηση από το νομικό σύμβουλο του Κοινοβουλίου και λάβαμε τη σαφή απάντηση της νομικής ε, επιτροπής του Κοινοβουλίου η οποία λέγει ότι το άρθρο 15 παράγραφο 3 και 4 προβλέπει σαφώς ότι πρέπει οι οργανισμοί να συμμετέχουν συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις για την πρόσβαση στα έγγραφα. Και είναι επίσης βασικό να τονίσουμε ότι ο εσωτερικός κανονισμός άρθρο 44 παράγραφος 4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι ε, ε, θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λαμβάνει ε, συγχρόνως τις προτάσεις που αναφέρονται ή στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στο εθνικό επίπεδο και τότε η Ευρωπαϊκή ε, το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να τα ε, ρυθμίζει συγχρόνως. Οπότε έχω παρουσιάσει τη θέση μου τώρα κύριε Πρόεδρε και την πρόταση της Νομικής Επιτροπής. Έχω διατυπώσει 53 τροπολογίες οι οποίες είναι στη διάθεση όλων Νομίζω ότι διατίθενται σε όλες τις γλώσσες και αναφερόμενος στην ε, δέσμευση που είχα αναλάβει έναντι της εκθέσεως Αργεντίνη και Χάουταλα ε, θα ε, επαναλάβω αυτό το οποίο έχουμε ήδη ψηφίσει δηλαδή να συσχετίσουμε τις δύο θέσεις αυτές εφόσον είναι συγγενή τα θέματα και οι 53 τροπο, από τις 53 τροπολογίες μας οι 43 ουσιαστικά εφαρμόζουν άμεσα τις τις συστάσεις της εκθέσεως Αργεντίνη. Ευχαριστώ όπως είπα την πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων οι οποίες με στήριξαν στην προσέγγιση μου. Βέβαια το ΕΛΚ δεν με στήριξε και ο σκιώδης εισηγητής τους έχει ανησυχίες τις οποίες δεν μπορώ να ικανοποιήσω αλλά κατά τα άλλα πιστεύω ότι ε, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στην έκθεση στις Αργεντίνη Χάουταλα και εις τις ε, τροπολογίες και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν υιοθετηθεί. Ευχαριστώ για τη σύντομη παρουσίασή σας και Προτού ακούσουμε τα σχόλια ε, της, ε, της ως συγητού ε, της κυρίας Σόμερ θα ήθελα να αναρωτήσω αν η Επιτροπή το Συμβούλιο θέλει να σχολιάσει και δίνει το λόγο στην Επιτροπή. Uh, Πολύ σύντομα. Η Κομισιόν διαφωνεί με την άποψη του σύγχυτη σχετικά με το άρθρο 15.3 της συνθήκης. Η δεύτερη πρόταση Κομισιόν σκοπεύει να εφαρμόσει το άρθρο 15.3 προσαρμόζοντας τον υφιστάμενο κονισμό στη συνθήκη της Λισαβόνας και αφήνοντας τη συζήτηση για τις λοιπές τροπολογίες ανοιχτή βάσει της πρότασης του 2008. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν θεωρεί ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε αμέσως τις ελέγξεις απαιτήσει της συνθήκης, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής του φυστάμενου κανονισμού και σε δεύτερο στάδιο να συζητήσουμε λοιπές τροπολογίες του κανονισμού για τον κανονισμό και αυτό είπε και ο κύριος Τσέπκοβιτς ε, σε σχέση με την έκθεση ΤΕΤΙΝΗ και επίση αυτό είναι το περιεχόμενο και τη επιστολή που έστειλε στη διάσκεψη των Προέδρων. Δεν θα ήθελα τώρα να σχολιάσω το περιεχόμενο των τροπολογιών αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Σχόλια από την Πολωνική Προεδρία υπάρχουν. Δεν θέλετε το λόγο μάλιστα. Παρακαλώ. Τα μέλη μπορούν να ζητήσουν το λόγο. Η κυρία Σόμερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να πω κάτι γιατί ο εισηγητής γράφει στην αιτιολογία της εκθέσεώς του ότι όλες οι ε, πολιτικές ομάδες συμφώνησαν η δεύτερη πρόταση να ενσωματωθεί στην πρώτη και να αποτελέσουν ένα σύνολο αλλά δεν είναι έτσι εμείς είπαμε ότι η δικιά μας προτεραιότητα είναι να προχωρήσει ε, ο κανονισμός όσο όσο πιο γρήγορα και να ευθυγραμμιστεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ε, ε, υπάρχει και κάτι διαφορετικό. Εμείς θεωρούμε ότι καταρχήν θα πρέπει να επεξεργαστούμε τη δεύτερη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε την πρώτη πρόταση μπορούμε να την επεξεργαστούμε σε το χρόνο. Οπότε ε, έτσι διεκπεραιώνω το καθήκον μου έναντι της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της ΑΦΚΟ που λέγει ότι οι δύο κανονισμοί είναι δύο, δύο παράλληλες νομοθετικές διαδικασίες ε, και είμαι πολύ επιφυλακτική παρόλες τις αξιολογήσεις των νομικών γιατί στη χώρα μας υπάρχει ένα ρητό ότι αν υπάρχουν ε, δύο νομικοί υπάρχουν πέντε γνώμες οπότε ε, μπορεί να υπάρχουν διαφορές ερμηνείας και απόψεως. Συμφωνώ με τον ε, ε, Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς ότι ε, η έκθεση Κάσμαν αναφέρεται σε πολλά θέματα που δεν έχουν άμεση σχέση με το δικαίωμα του κοινού να έχει πρόσβαση στα έγγραφα. Υπάρχει ένα μπέρδεμα και αυτό προβληματίζει την πολιτική μου ομάδα, ιδίως όσον αφορά τις διαθεσμικές συμφωνίες με το καθεστώς του Ευρωπαίου Ευρωπαίου διαμεσολαβιστή, δηλαδή δεν μπορούμε συλλήβδη να τα επεξεργαστούμε όλα αυτά σε αυτό το σχέδιο και επιπλέον αν κοιτάξουμε τα προβλήματα ανταγωνισμού και την προστασία των δεδομένων των ιδιωτικών επιχειρήσεων θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Υπάρχει αυτό που ονομάζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο intellectual property και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο μέλλον με τις δημοσιεύσεις διαβούλευσης για τις κοινοποιήσεις διότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λέγει ότι ζητούνται πάρα πολλά στοιχεία μεταξύ 10.000 και 15.000 σελίδων το οποίο είναι ίσως αξιοπερίεργο. Εδώ όμως δεν μιλάμε για την ποσότητα του κειμένου, για τον όγκο του, αλλά μάλλον ε, το περιεχόμενο και θα έπρεπε να βρεθεί μία λύση εκτός αυτού του του θέματος και να, να λάβουμε υπόψη μας και τη διαφάνεια για τον ε, ανταγωνισμό. Επίσης πιστεύω ότι η έκθεση έχει πολύ καλά στοιχεία, ποτέ δεν το αμφισβητήσαμε, αλλά ε, σε, η έκθεση αυτή κάπως ε, έχει περιοριστεί σε σχέση με την προηγούμενη και ουσιαστικά οι αλλαγές είναι διακοσμητικές. Το έχω ήδη αναφέρει στο στον εισηγητή και δεν θα πρέπει να με παρεξηγήσει. Θεωρώ όμως ότι το πιο βασικό είναι οι ορισμοί. Τι είναι τα έγγραφα, τι είναι οι αποφάσεις, τι είναι οι πληροφορίες. Όλα αυτά έχουν μείνει ακόμη πολύ ασαφή και επιπλέον υπάρχει απέτηση για, να, για μία πύλη ε, σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα, πράγμα το οποίο θεωρώ ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και εκφράζομαι εδώ πάρα πολύ προσεκτικά. Οπότε ουσιαστικά η έκθεση δεν άλλαξε και πολύ και πιστεύω ότι ο εισηγητής προσπαθεί να πιέσει το Συμβούλιο μέσα της δεύτερης εκθέσεως να διαπραγματευτεί μαζί του εφόλης της ύλης αλλά συνεχίζει να υφίσταται το νομικό κόλλημα εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία όσα αναφορά τα ε, ε, αρχικά στοιχεία. Ε, με την κυρία Χάουταλα είχαμε καταλήξει σε συμβιβαστικές λύσεις. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και πληροφόρηση της, του κοινού, αλλά δεν πρέπει να είναι άκρατη η πρόσβατη αυτή και επιπλέον υπάρχει το πρόβλημα της αναμίξεως των νομικών εγγράφων ε, διότι νομίζω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε την απόφαση ε, του ε, ε, ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και η δεύτερη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακριβώς συμμορφώνεται στις αποφάσεις αυτές. Οπότε ναι μεν θα συμφωνούσαμε στα συνταγματικά θέματα αλλά θεωρούμε ότι η δεύτερη πρόταση πρέπει να ρυθμιστεί κατά προτεραιότητα και να μην αναμειχθεί με τη διαδικασία του 2008. Δεν μπορώ εδώ να σας πω πώς θα καταλήξει το θέμα. Είναι θέμα πλειοψηφίας, δεν ξέρω αν θα παραπευθεί και πάλι στην Επιτροπή, αλλά θα δούμε πώς θα πάμε. Ευχαριστώ. Και τώρα αρχίζει η συζήτηση με την κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, αν και το θέμα νομίζω ότι πρέπει να πολυσυζητηθεί εδώ μέσα. Δέχομαι τη δουλειά του κυρίου Κάσμαν και συμμερίζομαι τους στόχους του. Τον διαβεβαιώνω ότι η Άλντε δέχεται πολλές από τις αλλαγές που προτείνει. Το θέμα που πρέπει να θέσουμε όλοι είναι σε ποιον ανήκουν αυτά τα έγγραφα εμείς οι σε εμάς τους ευρωβουλευτές, τους πολιτικούς γενικότερα ή στους δημοσίους υπαλλήλου της Ένωσης ή μήπως στους πολίτες, μήπως οι πολίτες είναι οι ιδιοκτήτες των εγγράφων αφού αυτούς αφορούν. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι για να αυξηθεί η διαφάνεια και με χαρά θα συνεργαστώ με τον κύριο Κάσμαν για να γίνουν μερικά παραπάνω βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα θα ασχοληθώ με ένα θέμα, τα δικαστήρια στο Λουξεμβούργο. Κατά τα πρώτα έτη της εφαρμογής αυτού του κανονισμού ήταν πολύ, είχαν πολύ διαφανή λειτουργία, μετά όμως φαίνεται ότι η διαφάνεια μειωνόταν. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Το δικαστήριο επέτρεψε στην Κομισιόν να θεωρήσει όταν χειρίζεται το θέμα της πρόσβασης στα έγγραφα, να θεωρήσει ότι εκείνη θα κρίνει όπως νομίζει. Δηλαδή, ότι εκείνη θα κατηγοριοποιήσει τα έγγραφα και επομένως τα θεσμικά όργανα μπορούν να θεωρούν ότι μόλις παραχθεί κάποιο έγγραφο είναι βασικά εμπιστευτικό. Αυτό αντιφάσκει με την νομοθεσία του 2001 και γι' αυτό δέχομαι την προτροπολογία του κυρίου Κάσμαν να διαγραφεί η πρόταση της Επιτροπής μερικά έγγραφα να εξαιρούνται από την νομοθεσία. Και νομίζω ότι πρέπει μάλιστα να είναι υποχρεωτικό για τα όργανα κάθε αίτηση να τη χειρίζονται μεμονωμένα. Ευχαριστώ. Ας σταματήσω εδώ αλλά θα συνεχίσουμε τη συνεννόηση. Φυσικά συμφωνούμε ότι το θέμα πρέπει να συζητηθεί. Αλλά ακριβώς αυτό γίνεται, συζητιέται, συζητιέται. Δεν είναι πρώτη φορά. Μάλιστα γι' αυτό ακριβώς η απόφαση και το τελευταίο ψήφισμα του Κοινοβουλίου κατέληξε σε αυτή τη δεύτερη εκδοχή της έκθεσης Κάσμαν. Θα συνεχίσει να συζητιέται λοιπόν ο κύριος Γιόγκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν είναι μόνο η κυρία Σάμερ σκιώδης, είμαι και εγώ για την ομάδα μου. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Λοιπόν, επί της ουσίας. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι συζητάμε γιατί αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές. Σε, όλα τα βαρόμετρα που βλέπουμε, τα ευρωβαρόμετρα, βλέπουμε ότι ο κόσμος αγνοεί όλο και περισσότερο την Ένωση, πράγμα που είναι άδικο. Και ορισμένες ομάδες πολιτών ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν περισσότερο, παίρνουν την πρωτοβουλία εκείνη, όχι οι Βρυξέλλες, κάνουν την προσπάθεια δηλαδή να ζητήσουν, να ρωτήσουν κάτι, αλλά συνήθως η Ένωση λέει δεν έχετε δικαίωμα πληροφόρησης γιατί είναι όλα εμπιστευτικά. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ. Και γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα με τον Μιχαήλ Κάσμαν. Είναι τόσο σημαντικό το θέμα που αν θέλουμε να γίνει η Ένωση κάτι, οτιδήποτε, πρέπει να είναι όσο πιο ανοιχτή γίνεται. Και έχει δίκιο επίσης και η κυρία Σόμερ ότι οι ορισμοί των πραγμάτων είναι πολύ δύσκολο να γίνουν, αλλά τουλάχιστον μερικοί από τους όρους που χρησιμοποιούνται εδώ ε, μπορεί να δημιουργήσουν παρεξηγήσεις που παρεμποδίζουν την πληροφόρηση των πολιτών. Πρέπει να συμφωνήσουμε επί των όρων αυτών όποιο θέλει μπορεί να καταθέσει τροπολογίες, αλλά γενικά φυσικά υποστηρίζουμε την έκθεση. Δύο άλλα θέματα τα έχω ξαναπεί σε προηγούμενες περιπτώσεις. Με ανησυχεί λίγο το θέμα του κόστους προς τον πολίτη, για τον πολίτη και το πρόβλημα ότι πρέπει να είναι κανείς στο ερώτημά του να έχει πάρα πολύ ακριβή διατύπωση αλλά δεν πρέπει να το κάνουμε τόσο δύσκολο για τον πολίτη να ζητήσει κάτι ακόμα και δεν ξέρει τον αριθμό του εγγράφου ή που ακριβώς βρίσκεται εμείς τα όργανα πρέπει να του δίνουμε αυτή την πληροφόρηση. Γενικά όμως επαναλαμβάνω και θα το ξαναπώ όπως το έχω ξαναπεί είμαι πολύ ικανοποιημένο από τη δουλειά του εισηγητή μας και του εύχομαι καλή επιτυχία στη συνέχεια. κυρία Αλφάνο είναι και αυτή σκιώδη για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κάσπαν για τη βαθιά του δέσπευση που και να εγγύθει τη διαφάνεια και την πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν κατορθώσουμε να βάλουμε τους πολίτες σε θέση να γνωρίζουν τι ακριβώς κάνουμε εμείς εδώ μέσα, τι κάνουμε, τι εγκρίνουμε, ποιους νόμους εγκρίνουμε και τι συζητάμε, δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία και επίσης ε, κινδυνεύουμε να συνεχίσουμε να χάνουμε την εκτίμηση των πολιτών και να αυξάνεται το κύμα κατά των πολιτικών ε, και πιστεύω ε, ότι δυστυχώς και η χαμηλή προσέλευση στις ευρωεκλογές ε, το δείχνουν αυτό. Ε, νομίζω ότι ε, για το να τοποθετηθούμε για τις δύο προτάσεις της Κομισιόν ταυτόχρονα ε, είναι κάτι καλό και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Εγώ είμαι η για την έκθεση για το οργανωμένο κλίμα στην Ευρώπη. Τον κρίναμε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο, στην Επιτροπή και αρκετές παράγραφοι και τροπολογίες αναφέρονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Εγώ θα στείλω και τροπολογίες ε, για να διασφαλίσω την ε, πνήρη ενεχνευσιμότητα της χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και νομίζω ότι η διαφάνεια και η πρόσβαση από τους πολίτες ε, στις νομοθετικές πράξεις είναι ένας καλός τρόπος για να ε, δείξουμε πώς ε, μπορούμε να λειτουργήσουμε προς το συμφέρον των πολιτών και πώς χρησιμοποιούμε τα χρήματα προς το συμφέρον των πολιτών. Έτσι λοιπόν, σε σχέση με την έκθεση αυτή υπάρχει η λοιπόν υποστήριξη των φιλελευθέρων. Η κυρία Ίντβελ, πριν να ξαναδώσουμε το λόγο στον κύριο Κάσμαν. Δύο σχόλια, Πρόεδρε. Καταρχήν, ε, η κυρία Ζόμερ είπε ότι δεν πρέπει να έχουμε περιόριστη πρόσβαση στα έγγραφα. Δεν νομίζω ότι κάποιο το πρότεινε αυτό. Γνωρίζουμε βέβαια από ε, από την ε, πράξη ότι έχουν καταχραστεί κυβερνήσει τους κανόνες για την πιστευτικότητα όχι για να προστατεύσουν κάποια ζωτικά συμφέροντα αλλά για να καλύψουν κάποια πράγματα που έκαναν και τι θα πρέπει να έχουν κάνει. Το είδαμε αυτό στην περίπτωση Παραδείγματο χάρη των απαγωγών τη Συρίας, δούμε και το Wikileaks. Ε, όλα όσα έχει κάνει το Wikileaks για ορισμένα θέματα που είχαν δηλωθεί απόρριτα, μπορεί να ήταν απόρριτα κάποια έγγραφα για πολύ καλου λόγου, αλλά ορισμένα ήταν απλώ για να καλυφθούν παράνομες δραστηριότητες λάθη των κυβερνήσεων. Δεύτερο, θα σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα που σχετίζεται και με το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Ξέρετε ότι έχουμε συνάψει μια συμφωνία με τους Αμερικανούς για τη διαβίβαση των τραπεζικών δεδομένων και πριν ε, την έναρξη των διαπραγματεύσεων, το νομικό τμήμα του Συμβουλίου εξέδωσε μια γνωμοδότηση σε σχέση με την καταλληλότητα έναρξης των διαπραγματεύσεων αυτών. Με το πόσο σκόπιμο ήταν το ότι υπήρξε αυτό το έγγραφο, μου τον έφεραν. Έτσι λοιπόν ζήτησα την δημοσίευση, δημόσια κυκλοφορία αυτού του εγγράφου, γιατί θεωρούσα ότι ήταν πάρα πολύ σχετικό με τη συμφωνία. Δεν ε, είχα πρόσβαση στο έγγραφο. Ούτε καν ε, ε, έφτασαμε στην ε, υπόσχεση δημοσίευση. Έτσι λοιπόν προσέφηκα στο δικαστήριο και η υπόθεση είναι ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τώρα. Ωραία. Οι κυβερνήσει μα είπαν αρχικά δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε το έγγραφο αυτό γιατί θα υπάρχει διαταραχή των διαπραγματεύσεων με τι ΗΠΑ και των σχέσεών μα με τι ΗΠΑ. Δεν μπορούμε λοιπόν να το δημοσιεύσουμε. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το επιχείρημα, αλλά Κατά ενδιαφέροντα τρόπο, τον προηγούμενο μήνα, όταν είχαμε μία ακρόαση για αυτήν την υπόθεση, το Συμβούλιο βρήκε και νέα δικαιολογία, νέα δικαιολογία λέει, και είπε ότι δεν μπορούμε να το δημοσιεύσουμε γιατί υπάρχει πρόταση για ένα ευρωπαϊκό PFTP και ένα ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθηση τη χρηματοδότηση τρομοκρατία και αυτό το έγγραφο είναι σχετικό λοιπόν και με αυτή την πρόταση. Έτσι λοιπόν πρέπει να είναι μυστικό το έγγραφο. Εγώ σαν δημοκρατία θα έλεγα ότι αν έχουμε πληροφορίε που είναι σχετικέ με τη συζήτηση για μια νομοθετική πρόταση, δεν θα πρέπει να είναι απόρριτε, αλλά θα πρέπει να είναι δημόσιε. Οι πολίτε έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν. Και πώ μπορούμε εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητούμε μια πρόταση τη Κομισιόν, αν οι σχετικέ πληροφορίε σκοπίμω μα αποκρύπτονται. Αυτό ε, είναι ένα ε, τρόπο που χρησιμοποιούνται οι κανόνε περί απορρίτου. Αυτό θέλω να πω στην κυρία Ζόμερ. Και νομίζω ότι αυτό συνιστά κατάχρηση των κανόνων. Ο κύριος Κάσμανος, ο συγητής. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, θα πρέπει να την τονίσω γιατί η κυρία Σόμερ ε, αναφέρθηκε στον διπρόεδρο Σεύκοβιτς. Ότι συμφωνεί μαζί του ότι οι τροπολογίες που χρησιμοποιώ στην τροπολογία μου πηγαίνουν παραπέρα εγώ θέλω να πω ότι ο κ. Σεύκοβιτ στην επιστολή του τη 26 Σεπτεμβρίου λέει, αναφέρεται στην προηγούμενη έκθεσή μου που επικαιροποιήθηκε Στη συνέχεια, έτσι λοιπόν, τα περισσότερα σημεία από τα οποία αναφερθήκε είναι τώρα ε, περτά και θα μπορούσε να έχει αναφερθεί στην εκθεσή μου που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο. Είναι δημόσια από την 1η Σεπτεμβρίου η έκθεση αυτή και Θέλω να σας πω, σε σχέση με αυτή την ε, λησβονοποίηση, δεν ε, είχαμε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το θέμα αυτό. Καμία απόφαση. Έτσι λοιπόν, ε, πρέπει το, το, πρέπει να το κάνουμε αυτό για να συμμορφωθούμε με κάποια απόφαση δεν είναι ορθό. Συμφωνώ με την κυρία Σομέρα στο εξή. Στο θέμα των νομικών γνωμοδοτήσεων. Δεν είμαι νομικός, αλλά Μία νομική γνωμοδότηση την λαμβάνω υπόψη, τη δέχομαι την απορρίπτω και πράττοντας αυτό επιλέγω και ε, το πολιτικό ε, τομέα. Δηλαδή αυτό ακριβώ κάνω εδώ πολιτικά. Είχα προετοιμαστεί να λάβω την απόφαση αυτή χωρίς να γνωρίζω αν θα με υποστήριζαν γιατί εδώ μιλάμε για πολιτική. Μιλάμε για ένα δικαίωμα το οποίο το ενισχύουμε. Σύμφωνα με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα περισσότερα ψηφίσματα που έχουν εγκριθεί από το δικό μας οίκο. Πολιτική είναι να το συμπεριλάβουμε αυτό στον κανονισμό και να προσπαθήσουμε, όπως είπαν και συνάδελφοι, να προσπαθήσουμε αυτή τη φορά και αυτή τη φορά περισσότερο από κάθε φορά πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Και πάλι στον κύριο Ντογιόν και στις Γερές να σας πω ότι αν ήμουν σαφή σε ορισμένα σημεία ευχαριστώ να συνεργαστώ μαζί σας για να πετύχουμε την διαφάνεια, τη σαφήνεια. Ξέρω ότι κάποια στιγμέ αποκλίνουμε από την ίδια προσέγγιση, αλλά ας ξεκινήσουμε λέγοντας τι μπορούμε να βελτιώσουμε με αυτό που παρουσίασα. Κυρία Σόμερ, δεν είπα στην αρχή ότι δεν αναφέρθηκα σε όλα τα πολιτικά κόμματα, είπα πλειοψηφία, ήμουν σαφής. Και αναφέρθηκα στο ότι και εσείς εκ μέρους ε, του ΕΛΚ ε, είχατε διατηρήσει κάποια απόσταση από τη δική μου προσέγγιση. Ήθελα λοιπόν ε, να είμαι σαφής γι' αυτό για να καταγραφεί. Τώρα, αν εξαναγκάζω το Συμβούλιο να διαπραγματευτεί, πολύ ωραία. Κάποιος πρέπει να το κάνει. Γιατί μέχρι τώρα δεν συμμετείχαν σε διαπραγμάτευση. Και δεν πρέπει να το ποτέ το τεκμήριο του απορρίτου. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε κατηγορίες εγγράφων. Πρέπει να εφαρμόσουμε τον κανονισμό. Και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 4, έτσι ώστε να εξετάσουμε ένα εγγραφό τη στιγμή την κατάλληλη, αν αυτό το έγγραφο δεν μπορεί να δημοσιευτεί, δεν μπορεί να αποκαλυφθεί στο κοινό γιατί υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις ή επειδή το γενικό συμφέρον δεν το επιτρέπει, πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό. Και δεν έχουμε τεκμήριο απορρίτου. Ευχαρίστως να, εργαστούμε, να εργαστώ στο θέμα των ορισμών. Δεν ε, πιστεύω και κάμε, αν ε, πετύχουμε μία συγκεκριμένη προσέγγιση, μπορούμε το χάρη να βάλει κάποιος πρόσβαση στα έγγραφα και μπορεί να ε, φτάσει κάποιος σε ένα μητρό που θα επιτρέπει στους πολίτες να το ερευνούν και να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες γιατί ε, ουσιαστικά δεν πετάμε τις πληροφορίες αυτού. Θέλουμε αυτοί να έχουν πρόσβαση, είτε μιλάμε για τις μη κυβερνητικέ την κοινωνία των πολιτών, οι πολίτες κτλ. Σύμφωνα με τη Σοφία για την εμπειρία της... σε σχέση με την πρόσβαση στα έγγραφα και σε συμφωνίες που αποτελούν ε, την βάση της νομοθεσίας και συχνά μας αρνούνται την πρόσβαση αυτή. Και να σας πω ότι το 2001 αν το Κοινοβούλιο δεν είχε βάλει στον αρχικό κανονισμό την ανάγκη για διοργανική συμφωνία σε σχέση με την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα έγγραφα, τότε πιθανότατα αυτή η διοργανική συμφωνία μπορεί ποτέ να μην είχε τεθεί σε ισχύ. Και να πω και κάτι ακόμα στην Κομισιόν. Έχω εργαστεί ε, με τον συνάδελφο για πάρα πολλά χρόνια και φυσικά το σεβούμε απόλυτα και τον εκτιμώ, αλλά θυμάμαι σε αυτή την επιτροπή, σε προηγούμενες τροπολογίες, όταν είχαμε συμπεριλάβει αναφορέ στην συνθήκη τη λειτουργίας τη Ευρωπαϊκής Ένωση, συγκεκριμένα στο άρθρο 15 και σε άλλα, όταν είχαμε τέτοιε παραπομπέ, μα είπαν ότι δεν ήταν απαραίτητες αυτές οι τροπολογίες, ότι το όλο θέμα τη Λισαβόνα. δεν θυμάμαι τον ακριβή όρο, αλλά θα ήταν κάτι σαν κομπέντιουμ. σαν επιτομή, αλλά αν ή ήταν τόσο σημαντική η λησβονοποίηση μέσα εισαγωγικά, γιατί η Κομισιόν περίμενε 18 μήνες, η ευθυγράμμιση δηλαδή με τη συνθήκη τη γιατί περίμενε η Κομισιόν 18 μήνε. Ήταν σαφέ ότι το Κοινοβούλιο θα ε, εξανάγκαζε το Συμβούλιο να διαπραγματευτεί. Γιατί θέλω να επενθυμίσω εδώ στους συναδέλφους ότι έχουμε εκλεγεί άμεσα για να κάνουμε αυτή τη δουλειά ως συνομοθέτες. Και δεν ε, θέλω να δεκτώ ότι ε, το κοινοβούλιο όποτε το βολεύει ακολουθεί την πολιτική των 27 κρατών μελών. Έχουμε ευρύ τομεί συνομοθεσία και θα πρέπει να συνομοθετούμε και να μην ε, αυτό νομοθετούμαστε. Και συγγνώμη αν παθιάζομαι εδώ, είναι μάλλον το μεσογειακό μου αίμα. Thank Σας ευχαριστούμε κύριε Κάσμαν. Έχουμε καθυστερήσει τώρα. Κύριε Σόμερ, ναι, αλλά πολύ σύντομα, ε. Γιατί έχουμε το τελευταίο σημείο και μετά τους συντονιστές. Συνεχώς καθυστερούμε και μετά έχουμε παράπονα. Βλέπετε τι ώρα είναι κύριε Πρόεδρε και τα λοιπά. Λοιπόν, παρακαλώ σύντομα, σύντομα. Είμαι σύντομα. Απλώς θα τα θέλω να τονίσω ότι το πρόβλημα δεν είναι εδώ να ε, ε, αποκρύψουμε έγγραφα από το κοινό γιατί ε, ζούμε σε δημοκρατίες με εκλεγμένους εκπροσώπους και στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει κανείς λοιπόν πρόσβαση στα έγγραφα της συνεδριάσεως και στο ίντερνετ μπορούμε να παρακολουθήσουμε από το διαδίκτυο δηλαδή οποιαδήποτε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το ξέρετε. Αλλά το πρόβλημά μου δεν είναι αν λέει μία συνάδελφο συνάδελφος από ο, τους φιλελευθέρους ότι δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη διαφορά των λόμπι ε, και εγώ θέλω να υπάρχει καταγραφή των λόμπι και νομίζω ότι πρέπει έτσι να ανταποκριθούμε ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του κοινού. Αλλά γενικώ και εμείς και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν πρέπει να θεωρούμε ότι αποκρύπτονται στοιχεία. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να διακηρύξουμε σαφώς και πρέπει να παραμείνουν στα χέρια των κρατών μελών. Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε αν θα αποκαλυφθούν ή όχι. Δεν μπορούν όλα να αποκαλυφθούν καλύπτονται. Παρακαλώ επιτρέψτε μου να το τονίσω αυτό. Είμαι υπέρ της ε, διαφανείας, μπορούν να γίνουν και παραπάνω πράγματα, αλλά πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την προσαρμογή στη συνθήκη της Λισαβόνας, χωρίς όμως ο ένας να κατηγορεί τον άλλον ότι ο ένας ε, είναι πιο πολύ υπέρ της διαφανείας και ο άλλος αποκρύπτει πράγματα. μια δημοκρατία γιατί αυτά δεν είναι επιτροπτά. Ευχαριστώ κυρία Ζόμερ. Μην ξαναξεκινήσουμε τη συζήτηση αλλά παρακαλώ θα ήθελα, εφόσον λέγεται στα πρακτικά ότι έχουμε το τελευταίο λόγο σαν εισηγητής, ε, εγώ άκουσα αυτά που είπε ο κύριος Κάσμαν, είπε η κυρία Ζόμερ και επανέρχομαι σε αυτό το οποίο είπα στην αρχή, ότι στο χέρι μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα άλλα θεσμικά όργανα θα διαπραγματευτούν μαζί μας. Σας ευχαριστώ που είσαστε σύντομα και τώρα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι 10 Οκτωβρίου τελειώνει η προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών και ε, θα πρέπει να ε, ψηφίσουμε τον Νοέμβριο και τώρα το επόμενο θέμα είναι για το TFTP ένα θέμα που θα μας παρουσιαστεί από τον κύριο Πρίμπε γρήγορα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης Χρηματοδότησης Ορμοκρατίας Διαθέσιμες Επιλογές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι συντομότερος από ό,τι είχα προβλέψει. Έχετε την ανακοίνωση μπροστά σας. Στόχος της είναι με βάση τις συζητήσεις που έγιναν στα πλαίσια της έγκρισης πέρυσι της συμφωνίας FTP και με τις προηγούμενες ανακοινώσεις να γίνει μια ενημέρωση. Λοιπόν, Αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή τη FTP είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε πώς και κατά πόσον μας χρειάζεται για να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία πανενωσιακός και πώς θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον αριθμό των ε, δεδομένων που παραδίδουμε σε τρίτες χώρες. Η πρόταση περιγράφει γενικά πώς θα μπορούσε να συνδεθεί το ευρωπαϊκό με το αμερικανικό σύστημα και ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις. Φυσικά συμπεριλαμβάνει, συζητάει και το κατά πόσον μπορεί να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και χρησιμοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερο υπαρχόντων συστημάτων. Η ανακοίνωση επίσης λέει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την απαραίτητη λιτότητα. Βέβαια δεν πρόκειται ένα τέτοιο σύστημα να είναι υπερβολικά ακριβό, αλλά θα χρειαστούν ορισμένοι πόροι. Και βέβαια άλλο βασικό θέμα είναι το εύρος τι περιορισμούς θα έχει το σύστημα αυτό στη χρήση παραδείγματος χάρη μόνο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή μήπως και γενικότερα καταπολέμησης εγκλήματος διαμεθοριακά. Και αυτό πρέπει να συζητηθεί. Επίσης είχαμε πει ότι τρεις εναλλακτικέ λύσεις υπάρχουν για να οικοδομηθεί ένα τέτοιο σύστημα. Αποκλείουμε μία καθαρά ενωσιακή όπως και μια καθαρά εθνική προσέγγιση και το κύριο θέμα που παραμένει μετά από όλα αυτά και με εσά φυσικά αλλά και με τα κράτη-μέλη είναι κατά πόσον όντως χρειάζεται ένα τέτοιο σύστημα. Χρειαζόμαστε ένα UTFTS πέρα από τις συμφωνίες που έχουμε με τρίτες χώρες. Εδώ πρόκειται για ένα πρώτο βήμα λοιπόν στην ανακοίνωση αυτή, δεν είναι τίποτε παραπάνω, δεν είναι πρόταση της Επιτροπής, ούτε προδικάζει το κατά πόσον πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα. Πρέπει να γίνει πρώτα αξιολόγηση και μετά να δούμε τι μπορεί ή δεν μπορεί να προτείνει η Κομισιόν. Η ανακοίνωση αυτή λοιπόν είναι μια πολύ πρώτη φάση συζήτησης όλων των θεμάτων που ε, τίθενται. Ευχαριστούμε κύριε Πρίμπε. Ήσασταν σύντομος και περιεκτικός. Ο κύριος Αλβάρο πρώτος, εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βέβαια ξέρω ότι έχουμε περιορισμένο χρόνο και θα ήθελα εδώ να επικεντρωθούμε σε λίγα σημεία καταρχήν με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Πήγε. Θα ήθελα να συμφωνήσω ότι είναι αναγκαίο αυτό το σύστημα αλλά πρέπει ο καθένας να έχει διαφορετική ε, διαφορετική αξιολόγηση και όχι αυτό το οποίο εμείς ίσως νομίζουμε διότι ε, παρόλη την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν νομίζω ότι το σύστημα λειτουργεί όπως θα έπρεπε ιδίως εάν κοιτάξουμε τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι έχουν κινήσει διαδικασία εδώ και ένα χρόνο και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν. Οπότε ήδη αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι δεν είναι ικανοποιητικό το σύστημα. Και η διαπίστωση αυτή ήταν διακομματική, δηλαδή ε, όλες οι πολιτικές ομάδες ε, συμφώνησαν ότι εμείς ε, είμαστε υπεύθυνοι για τα για τα στοιχεία των πολιτών μας ασχέτως του τι επιθυμούν οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ε, θέλω να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι αναγκαίο ε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ε, έχει ένα σύστημα δικό του για να συγκεντρώνει τα στοιχεία. Αλλά κανείς δεν έχει μιλήσει για ένα ευρωπαϊκό TFTP. Ίσως ορισμένες πολιτικές ομάδες το επιθυμούν, αλλά στο ψήφισμα σχετικά με τη συμφωνία TFTP και στο συνοδευτικό κείμενο κανείς δεν μιλά για το να έχει η Ευρώπη ένα ίδιο σύστημα και ε, θα ε, ήθελα να θεωρήσω ότι κανείς δεν το επιθυμεί εδώ που τα λέμε. Η οικονομική διάσταση ενός τέτοιου ο, συστήματος εφόσον πρόκειται για λογισμικό είναι ε, κάτι ανοιχτό γιατί ξέρουμε ότι το λογισμικό μπορεί να ε, έχει και προβλήματα. Πάντο συμφωνώ μαζί σας ότι ε, είναι βασικός ο τουρισμός αλλά πρέπει να καταπολεμήσουμε και την διασυροδιακή ε, εγκληματικότητα και ότι υπάρχουν σκοπιμότητες οι οποίες είναι πιο σημαντικές ίσως ε, από την προαναφερθήσα και ε, γι' αυτό βλέπω ότι υπάρχουν προσπάθειες ε, να παρουσιαστούν εδώ οι τρεις εναλλακτικές λύσεις και να προσεγγίσουν αυτό το οποίο επιθυμούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα είναι το πώς θα συγκεντρώνονται αυτά τα στοιχεία και εγώ θα ήθελα να ξέρω ποια θα είναι η νομική βάση. Θα είναι το άρθρο 16 και, ε, ή κάτι διαφορετικό. Σας ευχαριστώ για την ε, υπομονή σας. Τώρα όμως θα δώσουμε τον λόγο εις ε, του σκιώδη συγητή, στην κυρία Ζίμπελ και εγώ θα προσπαθήσω ε, να είμαι σύντομη και να εκφράσω μόνο ορισμένες ερωτήσεις. Με συνετάραξε η ερώτηση του κυρίου Πρίμπε ε, εάν το χρειαζόμαστε διότι για ορισμένου βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ήταν ο μόνος λόγος για τον οποίο επεκρότησαν την μέθοδο αυτή. Δηλαδή θα πρέπει εμείς να συγκεντρώνουμε τα στοιχεία μας διότι ε, γι' αυτό με ενοχλεί ότι ξεπερνούμε την εντολή. Ξεπερνά την εντολή Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχε ένα χρόνο για να παρουσιάσει μία πρόταση την οποία δεν έχουμε ακόμη και από την άλλη πλευρά συζητάμε πράγματα τα οποία ποτέ δεν θέλαμε να συζητήσουμε και τώρα ακούω ότι συζητείται επίσης αν θέλουμε να ασχοληθούμε μόνο στην έρευνά μας για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή για άλλα θέματα. Οπότε ε, δεν θα ήθελα όμως να ανοίξω μια τέτοια συζήτηση εδώ με αυτή την οδηγία. Τώρα χρειαζόμαστε ε, νέο, νέα περίπλοκη αρχή, νέο κτίριο, νέα συστήματα και αυτό θα μπορούσαμε ε, να λύσουμε με άλλο τρόπο. Η εταιρεία SWIFT ε, ε, διαμηνεί τα στοιχεία και η συγκέντρωση των στοιχείων μπορεί να οργανωθεί μόνο αν αυτό επιπτεύεται από τις ευρωπαϊκές αρχές. Πιστεύω όμως ότι το να απαλήφονται τα στοιχεία ε, ήταν ε, η μόνη προϋπόθεση την οποία είχαμε θέσει και τώρα πρέπει να βρούμε μία σύντομη λύση και να μην ανοίξουμε μία συζήτηση που δεν συμπεριλαμβανόταν εις ε, την εντολή. Ο κύριος Άλμπρεχτ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, διάβασα με πολύ ενδιαφέρον την ανακοίνωση αυτή και ο κύριος ο Πρίμπε άλλωστε μας είπε ότι η δημοσιονομική πλευρά είναι σημαντική και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Να αναρωτιέμαι λοιπόν αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια στιγμή θα σκεφτεί ε, ε, ε, και για ποιο λόγο καταρτίζει προγράμματα τα οποία δεν ζήτησε κανείς. Και το λέω αυτό σαφώς διότι βλέπω ότι υπάρχει μια, υπάρχει μια καμψία. Εμείς έχουμε πει σαφώς ότι δεν μας ενδιαφέρει ε, για ένα σύστημα σαν αυτό το οποίο έχουν οι Αμερικάνοι με το TFTP να αντιγράψουμε το ίδιο στην Ευρώπη και τα στοιχεία τα τραπεζικά για το SWIFT τα οποία διαθέτουμε σαν πακέτο δεν ε, πρέπει να θεωρηθούν σαν βάση για να υπάρξουν έρευνες. Δεν ήταν ποτέ αυτή η πρόθεσή μας θα μπορούσε να σταματήσει αυτή η μεταφορά στοιχεία εάν ε, δεν ικανοποιηθούμε σε αυτό που είπαμε. Δηλαδή ε, πως ε, όταν πρόκειται για στοιχεία που συγκεντρώνονται από το SWIFT μπορούμε να τα συγκεντρώσουμε αλλά σεβόμενοι την ομοθεσία και τα συνταγματικά δικαιώματα δικαιώματα και να αποφύγουμε την ε, μεσολάβηση τρίτων κατά περίπτωση. Θα μπορούσαμε ίσως να μεταδίδουμε ορισμένα τέτοια τραπεζικά συστήματα αλλά καλύτερα θα ήταν να μπορούμε να συγκεντρώνουμε όλα αυτά τα στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο κεντρικά και αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να εξεταστεί ε, αναλόγως των επιχειρήσεων και κατά περίπτωση αν υπάρχει ε, μία υπόνοια ή υποψία βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου διότι όταν εφαρμόσαμε τις διεθνές συμφωνίες δεν είπαμε πουθενά ότι θα προεξοφλήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική αλλά προσπαθήσαμε να συμμορφωθούμε στο αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης. Η κυρία προεξοφλησουμε την ευρωπαικη πολιτικη αλλα προσπαθησαμε να συμμορφωθουμε στο αποτελεσμα μιας διαπραγματευσης η κυρια Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι εδώ είναι το τελειότερο παράδειγμα ξεπλήματος πολιτικής που έχω ποτέ δει. Όπως είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι, κανείς δεν ζήτησε αυτό το σύστημα. Η Κομισιόν απλώς δεν έκανε, δεν εφάρμοσε αυτά που είχαν προβλεφθεί και αυτά που είχαν προβλεφθεί ήταν ότι η συμφωνία με τη ΣΥΠΑ θα εγκρινόταν μόνο με τον όρο μέσα σε ένα χρόνο να υπάρξει ένα σύστημα εξαγωγής στοιχείων, συλλογή στοιχείων. Είναι θέμα πολύ απλό, θέμα software, τίποτε παραπάνω. Δεν χρειάζεται καν ολόκληρος χρόνος για να δημιουργηθεί. Η πρόταση αυτή αφορά τη συλλογή και την αποθήκευση και τη διεκπαιρέωση στοιχείων μέσα στην Ευρώπη. Κάτι τελείως διαφορετικό δηλαδή. Εμείς δεν ζητήσαμε αυτό, ζητήσαμε και μας υποσχεθήκατε κάτι που δεν το πραγματοποιήσατε, δεν είστε α, εδώ εταίρος μας. Γιατί αν προτείνετε κάτι τέτοιο ξεπερνάτε ακόμη και αυτά που κάνουν οι Αμερικανοί. Δεν μιλήσατε για το SWIFT βέβαια, αλλά άμα διαβάσω την πρόταση καταλαβαίνω ότι καλύπτει και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ξεπερνάει ακόμη και αυτά που κάνουν οι Αμερικανοί με τα στοιχεία τους. Τέλος, νομίζω ότι είχατε έρθει όταν έθεσα προηγουμένως το θέμα της γνωμοδότησης του Συμβουλίου για τη συμφωνία με το SWIFT. Το ίδιο το Συμβούλιο θεωρεί στην προσφυγή του στο δικαστήριο ότι ακόμη και αν είχα ζητήσει να μην υπάρχουν τέτοια εμπιστευτικά έγγραφα πάλι θα το αρνούνταν το Συμβούλιο γιατί αφορά τη συζήτηση του θέματός σας. Αν όμως ισχύει αυτό κύριε Πρίμπε με ακούτε ή όχι. Δεν νομίζετε ότι θα ήταν φυσικό για μια δημοκρατία αν υπάρχει ένα έγγραφο για το οποίο το ίδιο το Συμβούλιο με την υποστήριξη της Κομισιόν θεωρεί ότι αφορά τη συζήτηση αυτή δεν θεωρείται ότι αυτό θα ήταν λόγος να δημοσιευτεί το έγγραφο μάλλον παρά να κρατηθεί απόρριτο. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να γίνει εδώ σοβαρή συζήτηση στο Κοινοβούλιο της πρότασής σας εάν διακρατάτε στοιχεία από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε κυρία Ιντφελτ. Τώρα, ευχαριστούμε τους διερμηνείς για τα πρόσθετα λεπτά που θα χρειαστούν για να απαντήσει ο κύριος Πρίμπε, χωρίς να τους το ζητήσουμε βέβαια. Τους ευχαριστούμε όμως. Ορίστε κύριε Πρίμπε μου όπως θέλετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά σημείωσα όλα όσα υπόθηκαν. Δεν ξέρω αν το θέμα του νομικού υποβάθρου έχει κανένα νόημα. Πια. Πάντως δεν έχουμε ακόμη αποφασίσει ούτε γι' αυτό. Μάλλον το 87 παρά το 60, αλλά δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Σημειώσαμε όμως όλα όσα είπατε. Υπάρχει και το 11, το σημείο 11 της συμφωνίας που μιλάει για τη δυνατότητα δημιουργίας ενός καινούργιου συστήματος, το οποίο είχατε δεχτεί κι εσείς. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες δυνατότητες υπάρχουν για τη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος. Για μας το πρώτο θέμα, ξαναλέω, είναι τι χρειάζεται σε ενωσιακό επίπεδο. Όχι πώς να καταργήσουμε τη συμφωνία Ένωσης είπα για, αυτό το, για ένα τέτοιο σύστημα, αλλά τι χρειάζεται από ευρωπαϊκής πλευράς. Και μετά να δούμε τι επιπτώσεις θα έχει ένα τέτοιο σύστημα σύμφωνα με αυτά που προβλέπει το άρθρο 11. Τα σημείωσα πάντως όλα όσα είπατε. Δεν έχω τίποτε να προσθέσω σε αυτή τη φάση. Σας κατευχαριστώ. Κυρία Ιντφελντ. Κοίταξτε, ως μέλος του Κοινοβουλίου βρίσκω απαράδεκτο να αρνείστε να απαντήσετε σε ερωτήματα. Δεύτερον, λέτε ότι δεν γνωρίζατε ότι το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει ένα σύστημα απλής εξαγωγής στοιχείων. Μα ακολουθήσατε ή όχι, δεν παρακολουθήσατε τις συζητήσεις του Κοινοβουλίου, ήσασταν παρόν σε όλες τις συζητήσεις. Διαβάστε τα πρακτικά. Αυτό που ζητήσαμε είναι σαφέστατο και εγώ θέλω απάντηση τώρα για το ερώτημα της ε, και κατάργησης του απόρριτου. Έχω ρωτήσει αυτό το πράγμα μπροστά στους συναδέλφους. Δεν είναι τόσο δύσκολο να απαντήσετε ναι, όχι. Δίνω το λόγο στον κύριο Πρίμπε. Με συγχωρείτε κύριε Άιντφελντ. Δεν σας άκουγα γιατί είχα ρωτούσα εδώ τους συναδέλφους σε ποιο έγγραφο ακριβώς αναφέρεστε. Αν μου το πείτε θα απαντήσω στο έγγραφο της προσφυγής. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το έχετε αυτό το έγγραφο. Είναι η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου του Ιουλίου 2009 πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τα ΣΥΠΑ. Κύριε Πρίμπε, πώς θέλετε τώρα να απαντήσετε. Όχι κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι σε θέση, αλλά θα επανέλθουμε για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση του κύριου Πρίμπε. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε τώρα παραπάνω. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρίμπε και νομίζω ότι θα πρέπει να περάσουμε στι συνεδρίε των συντονιστών. Κατανοώ την κατάσταση εδώ, αλλά ο κύριος Πρίμπε εδώ εκπροσωπεί την Κομισιόν και επιλέγει να πει αυτά που επιλέγει δεν μπορώ εγώ να τοποθετηθώ σε σχέση με το τι δεν επιλέγει να πει. Λοιπόν, προχωρούμε στην συνεδρία των συντονιστών και σας ευχαριστώ που θα παραπέρνατε στην αίθουσα όσοι έχετε το δικαίωμα να συμμετέχετε στη συνεδρία των συντονιστών. Και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας στις 9 το πρωί. Αύριο